και όλα αυτά μπορούμε να τα ε, ελέγξουμε στον αντίστοιχο ιστότοπο. Όπως γνωρίζετε συνεδριάσαμε την 3η 14 Ιουλίου, μια πολύ σημαντική μέρα για μας, τους Γάλλους. Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, με τους εκπροσώπους της Επιτροπής για μια διοργανική συνάντηση για τα θέματα των πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κατέθεσε μια λεπτομερέστατη έκθεση για τον χρονισμό των πληρωμών, μια έκθεση η οποία επιβεβαιώνει την κατάληξη του τριγωνικού διαλόγου για τις πληρωμές, ότι δηλαδή στο τέλος του 16 τα απλήρωτα στα πλαίσια του πολιετούς 7-13 δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα δύο δις. Με αφορμή αυτό είδαμε να έρχεται ε, και μία νέα έννοια στην επιφάνεια, τα λεγόμενα κρυφά υπόλοιπα. Είναι μία δυνατότητα η οποία δίδεται στην Επιτροπή όταν σαν παράδειγμα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για να ξεκινήσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στην προχρηματοδότηση καθυστερεί λίγο την απόφαση και η καθυστέρηση αυτή διευκολύνει λογιστικά θα έλεγε κανείς ε, και δεν φαίνεται το ποσό αυτό ε, στο ύψος των μη πληρωμένων υποχρεώσεων. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντα στις 14 Ιουλίου έγινε και συνάντηση ε, στην έδρα του Συμβουλίου του Τριγωνικού Διαλόγου για το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 όπως επίσης και για τον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2015, σύμφωνα πάντα με την εντολή της Ολομέλειας. Το Συμβούλιο ε, με αυτή την αφορμή παρουσίασε και την ανάγνωση που έγινε στο Κορεπέρ στις 9 Ιουλίου. Το Κορεπέρ αυτό προχώρησε σε περικοπές 575 ευρώ, εκατομμυρίων ευρώ, μείον 4% δηλαδή, και επίσης ε, οδηγήθηκε και σε μια μεγαλύτερη περικοπή στις πληρωμές κατά 1 δις 400 εκατομμύρια με πολύ σημαντικές ε, ε, περικοπές στους τίτλους 1 και 4, κάτι το οποίο ιδιαίτερα στο 1 είναι πρόκληση θα έλεγα, αν δει κανείς πως χρηματοδοτείται το Ταμείο Εγγυήσεων ε, για το ΕΦΣΥ. Το Συμβούλιο δικαιολόγησε τις περικοπές αυτές για τη μικρότερη δυνατότητα απορρόφησης και μικρότερο ποσοστό εκτέλεσης ενώ οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου επιβεβαίωσαν ότι οι ανάγκες αξιολογήθηκαν με πολύ σωστό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιδράσαμε σε αυτή την ανάγνωση και ο Χωσέ Μανουέλ θα μας πει περισσότερα σε λίγο. Η ανάλυση τώρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των πιλωτικών και προπαρασκευαστικών δράσεων είναι κάτι το οποίο παρουσιάστηκε με πολύ συνοπτικό τρόπο. Για τον προϋπολογισμό τώρα του 2015, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, έκτακτη. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα έχουν γίνει δεκτά. Θα το αξιολογήσει και η κυρία Γουαλιαζάμπαλ μετά. Ε, συζητήθηκαν και τα υπόλοιπα. Έγινε χθε μια συνάντηση με την λεγόμενη Τρόικα των Εξωτερικών Υπηρεσιών και ο κύριος Γκέγερ θα μας τα παρουσιάσει. Έγινε επίσης ε, και μια συνάντηση και ε, θα μας τα πει και ο κύριος Ντεπρέ που θα έρθει σε λίγο για το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επιμείνει στην εφαρμογή του άρθρου 27 της Διοργανικής Συμφωνίας. Το άρθρο 27 προβλέπει μία μείωση κατά 5% του προσωπικού των εξωτερικών υπηρεσιών μέχρι το 17. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι οι δύο, επί της αρχής, ε, επί αρχές επί των δημοσιονομικών θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στον τρόπο ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Αν και ο κύριος Ντεπρέ μας θύμισε ότι η τελευταία σειρά του άρθρου 17 αυτό το οποίο λέγει είναι ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές εκτός από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δηλαδή το 5% εφαρμόζεται υποχρεωτικά στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ για το Συμβούλιο, το οποίο το ίδιο έχει προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού από μόνο του, έχει πάντα μια διακριτική ευχέρεια ως προς αυτό, όπως και το Κοινοβούλιο. Όλοι ενθυμούμεθα την έκθεση του κυρίου Ντεπρέ ο κύριος Ντεπρέ δικαιολόγησε, τεκμηρίωσε το επίπεδο, τον αριθμό του προσωπικού μάλλον του Κοινοβουλίου. Αυτά τα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις να κάνετε γύρω από αυτό. Δεν το βλέπω. Συνεπώς θα δώσω χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τον λόγο στον εισηγητή μας, τον γενικό μας εισηγητή, γύρω από το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 16. Ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Φερναντές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνησε τις προτεραιότητες τις οποίες έχει ο προϋπολογισμός αυτός, τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες υιοθετήθηκαν στην Ολομέλεια έτσι κι αλλιώς και έχουμε πλέον την εντολή μιας ισχυρής πλειοψηφίας με ξεκάθαρες προτεραιότητες με δημοσιονομικές συνέπειες. Προάσπιση της απασχόλησης, προάσπιση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων και, της, και πρόθεση της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συνέπειες στην απασχόληση, έχουν συνέπειες όμως και στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Να μην ξεχνάμε ότι η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από την ανεργία στην Ευρώπη είναι οι νέοι. Τους νέους τους έχει χτυπήσει επίσης ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο είναι διπλάσιο από τις άλλες κατηγορίες. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν 6 δις για την περίοδο 14-20 που το 14-15 ήδη άρχισαν να δαπανώνται αλλά για το 16 δεν υπάρχουν χρήματα για νέες πρωτοβουλίες και γι' αυτό πιστεύουμε ότι το 2016 αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να υπάρξουν επαρχείς πιστώσεις για τη λειτουργία του προγράμματος αυτού. Θα ήταν ένα εξαιρετικά κακό μήνυμα να μην συνεχιστεί η διαδικασία. Από την άλλη, πάντα στον τομέα της απασχόλησης, τα προγράμματα τα οποία συνδέονται με αυτούς τους τρεις στόχους, ιδιαίτερα ε, με την τριπλέτα αυτή των στόχων, ε, αφορούν στο Horizon 2020, στο 1-1, και ε, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερα προσοχή ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρικιστούν οικονομικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την έννοια της εσωτερικής αλληλεγγύης. Όταν μιλάμε για εσωτερική αλληλεγγύη, η πολιτική συνοχή είναι αυτή η οποία έχει τον σημαντικότερο ρόλο. Και γι' αυτό λοιπόν τα μία όπως το κοινωνικό επιτρέπουν να βοηθηθούν οι ασθενέστεροι, οι φτωχότεροι, και θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι όλοι αυτοί, οι εμπλεκόμενοι, να γίνουν αντικείμενο φροντίδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν γίνει αυτό, αυτό θα έχει συνέπειες σε επίπεδο δημοσιονομικό. Έχουμε και άλλες εξωτερικές ε, θα έλεγα προκλήσεις όπως η μετανάστευση, η βοήθεια για την ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης και υπάρχει επίσης και άλλο ένα θέμα όπως η εσωτερική ασφάλεια. Όλα αυτά μου τα έδωσε σαν εντολή η Ολομέλεια για να προωθήσω το πολιτικό μας πρόγραμμα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου επίσης και για το ότι έχουμε στην διάθεσή μας ε, μια πρώτη ε, έγκριση, μάλλον συμφωνία καλύτερα από πλευράς της Προεδρίας θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία αντιμετωπίζει τις συζητήσεις μέχρι τώρα με ιδιαίτερο επικοδομητικό πνεύμα. Στα πλαίσια των προγραμμάτων και των βημάτων προόδου που έχουν μέχρι τώρα συντελεστεί στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου. Κάτι το οποίο θα έλεγα αλλάζει τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική διαδικασία. Ως Κοινοβούλιο λοιπόν ενωμένοι εμείς θα πρασπιστούμε τις προτεραιότητες μας έχοντας να αντιμετωπίσουμε όμως απέναντί μας τις προτεραιότητες του Συμβουλίου. Βλέπουμε ότι οι σαφέστατες σκληρές περικοπές του Συμβουλίου είναι απαράδεκτες, απαράδεκτες για τομείς όπως ε, οι υποχρεώσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση περαιτέρω και στις πληρωμές κατά ένα δις 400 εκατομμύρια παρά την άνεση που παρέχει το περιθώριο ιδιαίτερα στα πλαίσια της κατηγορίας 4 όπου 400, με 450 εκατομμύρια μειώθηκε και για το 1-1 υπήρξαν πάλι 400 εκατομμύρια μειώσεις, περικοπές. Πρόκειται για περικοπές προκλήσεις. Γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με το ΕΦΣΥ, με το λεγόμενο σχέδιο πρόγραμμα Juncker. Πάντα επίσης είπαμε ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 και το πρόγραμμα συνδέοντας ή διασυνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe, θα πρέπει να παραμείνουν αλόβητα από την εφαρμογή του ΕΦΣΥ και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην δημοσιονομική διαδικασία κανονικά. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να ανακτήσουμε τα ε, τα ποσά τα οποία έχουν περικοπεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Και στο Horizon 2020 υπάρχει μία σόρευση καθυστερημένων, κρυφών μη πληρωμών και γενικότερα καθυστερήσεων που ξεπερνάει το ένα δις. Με άλλα λόγια, ε, ναι μεν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε επίπεδο πληρωμών για το Horizon 2020, αλλά αυτό θα δημιουργηθεί ε, εφόσον υπάρξει περικοπή του 1 δις. Αυτό σημαίνει από την άλλη ότι έτσι και αλλιώς το Horizon 2020 έχει μια ιδιαίτερα υψηλή δυνατότητα εκτέλεσης και απορρόφησης χρησιμοποιούνται διαφορετικές παράμετροι για τον υπολογισμό των δύο αυτών κριτηρίων από πλευράς του Συμβουλίου. Οι κλίδες ανάγνωσης του Συμβουλίου είναι διαφορετικές. Εάν ακολουθήσουμε τη λογική του Συμβουλίου, το Horizon 2020 με υψηλά ποσοστά απορρόφησης και υψηλά ποσοστά εκτελεσιμότητας δεν θα πρέπει να τύχει περικοπών. Αλλά όπως είπα, στην πρώτη φάση του τριγωνικού διαλόγου γίνεται μια συνάντηση συζήτηση επί των γενικών γραμμών και επί αλγορίθμων μη κατανοητών, οπότε οι προτάσεις του Συμβουλίου είναι ε, ε, μη κατανοητές. Υπάρχει και το κόσμε, υπάρχει το Erasmus υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης. Ίσα ίσα διασώσαμε τις προτάσεις αυτές με τις βασικές περικοπές στο τέταρτο τμήμα. Στο Συμβούλιο τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν λειτουργεί το Συμβούλιο καλά. Αν πραγματικά μειώνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν καλό βαθμό εκτελεσιμότητας και απορρόφησης, αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός του Συμβουλίου κάνει εντελώς λάθος. 73 ε, εκατομμύρια ας πούμε για ε, Horizon 2020 στις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων ε, και ένα διπλάσιο περίπου ποσό στις πιστός πληρωμών είναι απαράδεκτο. Μειώνουμε ένα πρόγραμμα με πολύ καλές επιδόσεις ως προς την εκτελεσιμότητα και την απορροφητικότητα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να δοθεί ένα δις επιπλέον. Λοιπόν, σεβόμεθα τους στόχους τους οποίους έχουμε ήδη θέσει στα πλαίσια του Horizon 2020. Είναι στόχοι τους οποίους έχει υιοθετήσει και το Συμβούλιο και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και λογικοί σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα το Συμβούλιο. Το ίδιο γίνεται και με το μέσο Connecting Europe. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές μειώσεις ε, στον τομέα των πληρωμών. Λοιπόν, το Συμβούλιο λέγει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να επαναγράψει πιστώσεις οι οποίες έχουν περικοπεί στο παρελθόν. Νομίζω ότι στην ουσία αποφάσισαν να μειώσουν τα προγράμματα προδίδοντας την εμπιστοσύνη μας και ε, επιστρέφοντας σε ε, υπεσχημένα ενώ δεν θα έπρεπε αυτό γιατί φύγουν όπως είπα προγράμματα με υψηλά επίπεδα απορροφητικότητας και εκτελεσιμότητας. Όσον αφορά το εργαλείο για την γειτονία, είχαμε περικοπή 103 εκατομμύρια και όσον αφορά την μείωση της στόχιας και το κεφάλαιο του σχετικό, που στηρίζει την αλληλεγγύη, το στόχο για την αλληλεγγύη και εκεί έχουμε μια περικοπή 50 εκατομμυρίων. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και στις περιοχές αυτές της Ευρώπης και στην γειτονιά της Ευρώπης, την κοντινή. Είχαμε περικοπή λοιπόν στα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί και διατίθενται για μετανάστευση για το άσυλο. Στο άσυλο έχουμε περικοπή 5 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό είναι σε αντίθεση με τις ε, αποφάσεις που έχει λάβει το Συμβούλιο. να, να μην αναφέρω και τη δική μας θέση. Λοιπόν, για το κατηγορία 1β, στα κονδύλια αυτά που επέτρεπαν την ολοκλήρωση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει και τις υποχρεώσεις που έχουμε όσον αφορά τις πληρωμές. Έχουμε ε, συνάψει μια συμφωνία, υπάρχει διοργανική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ούτω ώστε το 2017 να μην υπάρχουν ε, δύο δις ευρώ σε μη πληρωμές όσον αφορά τα προγράμματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τα προγράμματα που έταξαν στην περίοδο 2007 μέχρι 2013. Η κατάσταση λοιπόν θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτη από πλευράς του Συμβουλίου διότι βασιζόμαστε σε μία αρχή την αρχή του σεβασμού των υποχρεώσεων, των ανηλυμένων υποχρεώσεων και ο σεβασμός των ανηλυμένων υποχρεώσεων σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να σεβόμαστε μόνο τις ανηλυμένες υποχρεώσεις φάση πληρωμές αλλά και αυτά που προβλέπονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε υιοθετήσει στοιχεία χαμηλότερα από εσά περίοδο 2000 μέχρι 2013 χρησιμοποιώντας το εργαλείο ευελιξίας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέσο ευελιξίας και στο πολιετές πλαίσιο. Και αυτό μας θυμίζει ότι έχουμε ελάχιστα περιθώρια στα διάφορα κεφάλαια. Στο, στην κατηγορία 3 δεν έχουμε ε, κανένα περιθώριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται κατώτερα, σε κατώ, με κατώτερα ποσά να μην χρησιμοποιούμε το μέσο ευελιξίας. Πρέπει όμως να το χρησιμοποιούμε το μέσο ευελιξίας για την κατηγορία 3 και για τις άλλες κατηγορίες. Παραδείγματο χάρη για την 1α όπου θέλουμε να συνεχίσουμε κάποιες πρωτοβουλίες και για την 1Β όπου θέλουμε να συνεχίσουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων όπως ε, υπενθύμησα. Ιδού λοιπόν αυτή είναι η θέση μας. Λοιπόν το μέσο ευελιξίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για την κατηγορία 3 αλλά και τις άλλες κατηγορίες να μην λησμονούμε ότι η ευελιξία εδράζεται επί μιας νέας ενίας, μιας ενίας που ήδη χρησιμοποιήθηκε και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων ε, που καλείται σχέδιο Juncker. Έχουμε ένα περιθώριο γενικό ε, που ξεκινάει από το 2016. Τι σημαίνει αυτό το περιθώριο, το γενικό. Σημαίνει ότι το περιθώριο των υποχρεώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τα προηγούμενα χρόνια μπαίνει σε ένα γενικό απόθεμα και αυτό το γενικό αποθεματικό ε, μπορεί να χρησιμοποιείται για στόχους πολιτικούς ειδικού συγκεκριμένους. Σημαίνει για την ανάπτυξη, για την απασχόληση μεταξύ άλλων και πιο συγκεκριμένα για την απασχόληση των νέων. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο ευελιξίας, μέσω ευελιξίας, μια ευελιξία που δεν πρέπει να λησμονεί το Συμβούλιο και θέλουμε αυτό το μέσο να χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να επιθυμίσουμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι μικρό προπολογισμό, είναι 1% του ΑΕΠ ε, και πλαισιώνεται σε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μας παρουσιάζεται ένας προπολογισμό με μειώσεις. Μειώνει έτσι περαιτέρω το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το Συμβούλιο και αυτό που βρίσκουμε στο πλαίσιο είναι μειωμένο. Έτσι δε περαιτέρω τα στοιχεία που παρουσιάζονται περισσότερο, λιγότερα τα ποσά από αυτά παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα παράδοξο. Όλο ο κόσμο ξέρει ότι ομόφωνα υιοθετήθηκε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εν συνεχεία πώς κάποια κράτη-μέλη που καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ τα, οι αριθμοί είναι χαμηλότεροι από αυτούς που είχαν προγραμματιστεί στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που συστηματικά καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί προηγουμένως στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επανεντάξουμε να αποκαταστήσουμε τους αριθμούς που έχουν μειωθεί, τα ποσά που έχουν μειωθεί από το Συμβούλιο και να έχουμε τα κατάλληλα ποσά για να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις. Είναι σαφής η θέση μας, είναι ενωμένο το Κοινοβούλιο, έχουμε προτεραιότητες που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες και αν η συνεχεία χρειαστεί θα μπορούσα να σας δείξω ποιες μειώσεις παρουσιάστηκαν κατά κατηγορίες και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά αυτές οι μειώσεις είναι σε αντίθεση με τις θέσεις μας και με τις θέσεις του Συμβουλίου και θα βοηθήσουμε το Συμβούλιο ε, να μην αυτοπυροβοληθεί και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μία συνοχή όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Γενική Συγκητά. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν για μία αντιπαράθεση δύσκολη. Αλλά είπατε στο τέλος ότι έχουμε έναν πρόεδρο του Συμβουλίου ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός, ε, αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες μας ίσως συνδέεται και με την κεκτημένη εμπειρία της Λουξεμβουργιανής ε, Προεδρίας που έχει επιφορτιστεί με τη 14η Προεδρία του Συμβουλίου. Ο κ. Γκεγέρ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνούμε με τον συνάδελφο Φερνάντες. στα βασικά σημεία. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τις εκτιμήσεις του να κάνω κάποιες συμπληρώσεις. Εάν υπάρχει κάποια μέθοδος ε, στον τρόπο εργασίας του Συμβουλίου, δεν υποστηρίζω, απλώς τον ε, περιγράφω. Ασχολούνται μόνο με όσα σημεία του προϋπολογισμού προτείνει να αυξηθεί η Κομισιόν από χρόνο σε χρόνο και τα περικόπτουν. Ο δεύτερος τομέας όπου φαίνεται πώς δρά το Συμβούλιο είναι ότι θεωρούν ότι ορισμένα προγράμματα δεν απορροφώνται επαρκώς και εδώ κάνουν επίσης περικοπές. Μπορεί έχουμε, να έχουμε εμείς άλλη εκτίμηση για το γιατί υπάρχει αυτό το ποσοστό απορρόφησης <clears throat> και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για διάφορα θέματα μέσω διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω συζητήσει με εκπροσώπους του Συμβουλίου και ασχολήθηκα, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με την περιφερειακή πολιτική, με τις περικοπές σε διάφορα σημεία της περιφερειακής πολιτικής. Και η απάντηση του Συμβουλίου είναι ότι καθυστερούν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες, σε κάποια μεγάλα κράτη-μέλη ιδίω, να υποβάλουν προτάσεις για προγράμματα. Οπότε θεωρούν ότι θα υπάρξει χαμηλότερη απορρόφηση στην κατηγορία αυτή από ό,τι θέλουμε και εμείς και το Συμβούλιο. Παρά το ότι μπορεί να συμφωνούμε για τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σωστές προτεραιότητες που ανέφερε ο συνάδελφος Φερνάντες, θα είχε έννοια να δούμε εάν σε κάποια σημεία της περιφερειακής πολιτικής ε, τα κονδύλια είναι υπερβολικά. Θα μπορούσαμε δηλαδή από εκεί να πάρουμε κονδύλια για άλλα σημεία που χρειάζονται αυξήσεις. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Γιατί το σχέδιο προϋπολογισμού δεν μας λέει πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της χορήγησης επαρκούς χρηματοδότησης στο ΕΦΣΥ. Να υπενθυμίσω. Θεωρήσαμε ότι είναι καλό που πέρασε το ΕΦΣΥ, αλλά αν δούμε το χρηματοδοτικό του τμήμα, την πρικοδότησή του δηλαδή, ότι λέμε ότι θα πάρουμε μέχρι το 2020 από το περιθώριο 3 αντί για 2 δις, οπότε 5 δις πρέπει να βρεθούν από τους τρέχοντες προϋπολογισμούς. Έχουμε περικοπές ε, στο συνδέοντα στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Παρόλα αυτά, πρέπει να βρούμε αυτά τα 5 δις. Και ξέρουμε ότι Υπάρχει πολύ περιορισμένο περιθώριο, πολύ περιορισμένα διαθέσιμα μέσα, διαθέσιμες πιστώσεις για να βρούμε αυτό το, τα πέντε δις εκτός εάν κατά την ε, αναθεώρηση των πολιτών προοπτικών γίνουν ε, οι αναγκαίες μεταφορές πιστώσεων. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν θα ήθελα να βασιστούμε εκεί. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμεθα με το Συμβούλιο για να δούμε πού θα βρούμε αυτά τα πέντε δις και τα επιχειρήματά μας πρέπει να είναι τα επιχειρήματά μας πρέπει να είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και να ανταποκριθούν στα αιτήματα του Κοινοβουλίου χωρίς να περικόψουν περαιτέρω όμως ε, το συνδέοντας την Ευρώπη και τον ορίζοντα 20, 2020. Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα ήθελα εδώ να μου δώσετε τη γνώμη σας. Θα ήθελα να μου πείτε επίσης πώς μπορούμε να βρούμε άλλες χρηματοδοτικές ε, μεθόδους που να μοιάζουν με την πολιτική χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ να δούμε εάν θα μπορούσαμε αυτά τα νέα μέσα να τα συνδέσουμε με τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Αυτό θα ήταν μια ιδέα. Μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εξάλλου για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για αυτήν καταδεικνύει ότι αυτά τα μέσα που στις τελευταίες ε, προοπτικές παρουσιάστηκαν σαν η νέα πανάκια για τη χρηματοδότηση, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργούν τόσο καλά. Τώρα για τους νέους κανονισμούς που ισχύουν για το 14-20 θα λειτουργήσουν καλύτερα, θα το δούμε. Να δούμε λοιπόν τα χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς ε, η χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μεταξύ μας. Η Κομισιόν, δεν περιμένω βέβαια τώρα αμέσω, είναι σημαντικό όμως η Κομισιόν για την απόφαση το Σεπτέμβρη να μας πει η Κομισιόν πώς εκτιμά το ποσοστό απορρόφησης στα βασικά προγράμματα που έχουν περικοπεί από το Συμβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Τώρα για τους ε, εξωτερικούς φορείς. Ε, αυτοί απορροφούν ε, λιγότερο από 1% του προπολογισμού. Άρα δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επίμαχο θέμα. Οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο είναι περιορισμένες, μετριοπαθείς. Παίζουν όλο βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν είναι λογικές. κάνουν περικοπές 5.000 ε, στους προπολογισμού ε, κάποιου εξωτερικού φορέα. Τι ε, επίπτωση θα έχουν τέτοιες περικοπές. Ρώτησα, δεν μου απαντήσανε. Γιατί τις κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η καλή εκτέλεση του προπολογισμού και δεν μου έχουν απαντήσει, επαναλαμβάνω. Το πρόβλημα είναι το προσωπικό για αυτούς, του εξωτερικούς, για αυτούς τους εξωτερικούς φορείς. Το είπαμε και χθες όταν ακούσαμε την τρόικα των ε, φορέων που ήταν χθε εδώ. Έχουμε ήδη αποφασίσει ένα προϋπολογισμό που προβλέπει ενίσχυση της πολιτικής ε, μετανάστευσης, για παράδειγμα αύξηση θέσεων για την Europol. Και τώρα βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός ε, του 2016 της καταργεί. Τι προγραμματισμός είναι αυτός πολιτικής. Εκεί που λέμε ότι πρέπει οι εξωτερικοί φορείς να μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, αυτό πρέπει να εκφράζεται και στο οργανόγραμμα των φορέων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σόλμπριχτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τα πολωνικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ στο ζωζέ και θα ήθελα να εστιαστώ επί μίας πτυχής τη περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αναλύσει την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και έτσι έχουμε μεταφέρει χρήματα από το 2014 προς το 2015 διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποια επιχειρησιακά προγράμματα. Ήδη σήμερα έχουμε εγκρίνει περίπου τα μισά επιχειρησιακά προγράμματα. Είμαστε στο δεύτερο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών. Έχουν εγκριθεί πάνω από 300 επιχειρησιακά ε, προγράμματα και το ερώτημα είναι γιατί έχει ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση. Η μη έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων οφείλεται στα κράτη-μέλη ή σχετίζεται με κάποιες καθυστερήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πόρους ε, για μελλοντικά έτη. Ήδη το έχουμε κάνει. Πρέπει να το εξετάσουμε. Αν έχουμε πόρους για την περιφερειακή πολιτική, από αυτά που μας είπε ο συγητής, σημαίνει ότι έχουμε δύο κονδύλια στην πολιτική συνοχή, ένα από, για τα παλιά προγράμματα και ένα κονδύλι για τα νέα προγράμματα. Αν τα νέα προγράμματα δεν είναι έτοιμα, μπορούμε τελικά να χρησιμοποιήσουμε πόρους για να καλύψουμε τις καθυστερήσεις. Διότι φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε πόρους για να καλύψουμε κενά που υπάρχουν, αλλά αν υπάρχουν και άλλοι πόροι, τους περικόπτουμε αντί να καλύψουμε τις καθυστερήσεις. Αν δεν έχουμε ακόμα νέα προγράμματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του διαθέσιμους για να καλύψουμε καθυστερήσεις στην εκτέλεση προγραμμάτων. Και έτσι ε, μειώνουμε γενικά τα προβλήματα με τη μεταφορά των πόρων. Δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Και ρωτώ τον εισηγητή, Ποιε είναι οι συνέπειες για τον προπολογισμό για το 2016 έχουμε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δόθηκαν χτε. μα ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια άλλη αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες περί περιφερειακή πολιτικής για την Ελλάδα. Μεγαλύτερε προκαταβολές το 2016, άλλο ένα 5% και στήριξη μέχρι 100% στα προγράμματα για την περίοδο 2007-2013. Αυτό σημαίνει περισσότερους πόρους για την πολιτική συνοχής. Και ρωτώ, πώς σχετίζεται αυτό, πώς τα δύο πράγματα αυτά σχετίζονται, ποια η σχέση μεταξύ τους, αύξηση και μείωση ταυτόχρονα. Σίγουρα την καθυστέρηση όσον αφορά τα προγράμματα είναι κάτι που διευκολύνει την ε, καλύψη των μη πληρωθέντων ποσών. Τι θα γίνει όμως στην περίοδο 2017 μέχρι 20. Θα έχουμε έκρηξη των αναγκών και σίγουρα θα έχουμε πολλούς απλήρωτους λογαριασμούς. Όσον αφορά την Ελλάδα φυσικά θα υπάρξει ε, αντίκτυπος όσον αφορά το επίπεδο των πληρωμών. Ο κύριος Ντονάνο. Ευχαριστώ. Όπως και πολλοί άλλοι γενικά συμφωνώ με τους προσανατολισμούς του Γενικού Εισηγητή κ. Φερνάντες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, απασχόληση των νέων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό να μην το ξεχάσουμε. Και το θέμα της εξωτερικής αλληλεγγύης και για πολλά άλλα συμφωνώ. Θέλω όμως να επιμείνω στο γεωργικό θέμα. Χθες βράδυ υπέβαλα στην Επιτροπή Γεωργίας το σχέδιο γνωμοδότησής μου και η Επιτροπή με παρακάλεσε να ζητήσω να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των μέτρων για την στήριξη της αγοράς. Έχουμε πρόβλημα με τον γαλακτοκομικό τομέα, έχουμε κρίσεις υγειονομικές, ίσως και κλιματικές κρίσεις, έχουμε το πρόβλημα της Ουκρανίας. Άρα υπάρχουν πολλές ανησυχίες μεταξύ του κόσμου της υπαίθρου και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αξιοποιήσουμε όλα τα περιθώρια μέχρι το ανώτοτο όριο. Είναι εντελώς απαράδεκτο να μην ε, αξιοποιούμε πλήρως ε, τα περιθώρια του πολιετούς πλαισίου. Ανησυχώ πολύ, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή Γεωργίας ομόφωνα ζήτησε λοιπόν να αντισταθούμε στο Συμβούλιο, να επιβάλλουμε ένα προϋπολογισμό που να είναι καλύτερος από αυτόν που μας έχει υποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όπως έλεγα. Ευχαριστώ τον εισηγητή ο οποίος ε, παρουσίασε με μεγάλη ακρίβεια την κατάσταση πραγμάτων και διαρωτώ με κι εγώ γιατί το Συμβούλιο επιβάλλει αυτές τις περικοπές και μάλιστα σε σημαντικούς τομείς. Για παράδειγμα το κόσμο, την ε, πολιτική μετανάστευση, το έρασμο συν και για άλλα προγράμματα. Πρέπει πραγματικά να θέσουμε τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο. Πού οφείλονται, ποια είναι τα αίτια για αυτές τις περικοπές. Και τίθεται το ερώτημα ακριβώς εάν αποτιμώνται σωστά και ρεαλιστικά αυτά τα προγράμματα, αν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Πού πάνε αυτά τα κονδύλια που περικόπτονται, δηλαδή αυτά τα ποσά που περικόπτονται, γιατί υποθέτω ότι πάνε σε άλλα προγράμματα. Επίσης έχουμε το θέμα των καινοτόμων επιχειρήσεων που, επιχειρήσεων που εισάγουν καινοτόμα τεχνολογία. Και αυτές πρέπει να υποστηριχθούν ασχολούμεθα επαρκώς με αυτές. Τις πλαισιώνουμε με την προσοχή που χρειάζονται όταν εκινούν, όταν είναι startup. Πολύ συχνά ε, διαπιστώνουμε ότι αυτά τα startup που έχουν ε, πολλές προοπτικές, εισάγουν ε, πολύ σημαντική νέα τεχνολογία, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς από τι τράπεζε και άλλους ε, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και πολλές φορές εγκαταλείπουν την προσπάθεια και για το μέλλον της Ευρώπης οι επιχειρήσει αυτές είναι πολύ σημαντικές. Ίσως δεν έχουμε επαρκώς καλό διάλογο με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά στο μέλλον. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα με το Συμβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Σολίνη. Για το θέμα αυτό, χθε είχαμε ένα πολύ ενδιαφέροντα διάλογο σε μια ακρόαση για τη χρηματοδότηση των καινοτόμων επιχειρήσεων ακριβώ. Και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Η κυρία Τόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να στηρίξω τον Γενικό Εισηγητή Τελικά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε περικοπές τέτοιου είδους παρά ένα πολιετές δημοσιονομικό ήδη μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Και να πω επίσης ότι τελικά φτάνουμε στα όρια. Φτάνουμε στα όρια τα οποία πλέον δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της πολιτικής συνοχής, το πρόβλημα της καθυστέρησης της πιστοποίησης των προγραμμάτων, γιατί εδώ υπάρχει μεν ευθύνη των κρατών μελών, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όμως και το λέγω και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, Έχουμε στην καλύτερη περίπτωση μία προσπάθεια μείωσης των, του κόστους και μία προσπάθεια ταυτόχρονα με έμεσο τρόπο μείωσης του ίδιου του προϋπολογισμού. Γιατί ε, με τις συνεχείς αναβολές ε, κερδίζουμε λογιστικά. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα εδώ ε, των απλήρωτων λογαριασμών, κάτι το οποίο συμμετέχει και αυτό ουσιαστικά στη μείωση του προϋπολογισμού. Αυτό ισχύει όπως είπε και ο Ντενανό και για την Επιτροπή Γεωργίας. Εγώ ήμουνα στην Επιτροπή Αλίας. Η ίδια διαπίστωση, η ίδια αγανάκτηση για τις περικοπές, για έναν ελάχιστο προϋπολογισμό. θα πρέπει να πούμε ότι το Συμβούλιο στην παρούσα φάση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πολιτικών της σε επίπεδο δημοσιονομικό. Ε, ε ξέρουμε ότι το πρόγραμμα Juncker σαν παράδειγμα, οι πολιτικές της συνοχής και με την προσθήκη που αφορά την Ελλάδα, ε, τα θέματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας είναι θέματα τα οποία συμφωνούμε, στα οποία συμφωνούμε όλοι πολιτικά, αλλά σε επίπεδο δημοσιονομικό δεν παίρνουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Λοιπόν, πέραν του διαλόγου, πέραν των συμφωνιών και συζητήσεων, εμείς σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών με φωνή πιο δυνατή από ό,τι στο παρελθόν, να καταγγείλουμε την διπλή γλώσσα του Συμβουλίου. Αναλαμβάνει πολιτικές υποχρεώσεις το Συμβούλιο που δεν ακολουθούνται από υποχρεώσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού, σε επίπεδο δημοσιονομικό. Λοιπόν, φτάνουμε τα όρια μας. Νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει πέρυσι στα όρια μας, αλλά δυστυχώς οι δυσκολίες συνεχίζονται και δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε μόνο μέσω του διαλόγου με το Συμβούλιο. Είναι δυσκολίες ε, οι οποίες ε, θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστούν ίσως και μέσω καταγγελίας αυτής της έλλειψης ευθύνης, της διαφοράς ανάμεσα στις υποσχέσεις και στις ευθύνες. Yeah. Eh, I want to thank Fernandez for the Ευχαριστώ τον κύριο Φερνάντε. Μα και γράψε πολύ καλά την κατάσταση. Δεν θα επαναλάβω τα υποθέτα. Όλοι είμαστε συντονισμένοι. Έχουμε καθήκον να δούμε πώ μπορούμε να είμαστε κοινωνικά πιο προοδευτικοί. Ανεφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στην Ιρλανδία έχουμε τεράστια ζητήματα, όπω και άλλε χώρε με τα θέματα τη αλληλεία και τη γεωργία. Η αλληλεία και η γεωργία είναι βασική πηγή τη οικονομία και θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να διαφυλάξουμε του τομεί αυτού και κυρίω ε, την πρωτοβουλία για την ενεργεία των νέων αυτό αφορά την Ευρώπη και βλέπουμε ότι οι νέοι μας είναι οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί από την κρίση. Εγώ θα στήριζα οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει δυνατότητες προχρηματοδότησης, κυρίως ε, άμα μιλάμε για τα προγράμματα εκείνα, στα οποία φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ε, μικρή. Γιατί υπάρχει ε, αυτό το πρόβλημα και πώς βλέπουμε το λόγο της κατανομής, πώς κατανέμονται οι πόροι στα κάτι μέλη για τις χώρες που δεν έχουν τους πόρους. Μπορούμε να τα επαναξετάσουμε όλα αυτά. Πέραν αυτού, κύριε Φερνάντες, έχετε την ευρία υποστήριξη του Κοινοβουλίου, όπως είπατε. Και ελπίζω τελικά να καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερνάντες, αν έχει την καλοσύνη, να ολοκληρώσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Μαραγκάλ. Ο Μαραγκάλ πρώτα. Ευχαριστώ. Μόνο ένα σχόλιο γενικό. Άκουσα την παρουσίαση του κυρίου Φερνάντες, πολύ σαφή, πολύ συγκεκριμένη, για το τι μπορούμε να περιμένουμε για αυτόν τον προϋπολογισμό και τη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Λοιπόν, για μένα ένα πόρισμα. Υπάρχει μια ευρεία συμμαχία στο σώμα μας που είναι λογικό να υπάρχει διότι ορισμένες ομάδες είναι ευρωσκεπτικιστικές. Είναι παρούσες εδώ και έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν αυτή την άποψη. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι και οι πραγματικοί ευρωσκεπτικιστές όμως είναι αλλού. Είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι οι πραγματικοί ευρωσκεπτικιστές. Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός είναι το βασικό μέσο λειτουργίας κάθε δημόσιου φορέα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ελάχιστη εμπιστοσύνη σε κάθε δημόσιο φορέα. Αυτοί εμποδίζουν την Ευρώπη να λειτουργήσει. Πρέπει να το πούμε αυτό γιατί είναι προφανές. Εντάξει, προσπαθούμε να βελτιώσουμε κατά 0,1 το ένα, 0,2 το άλλο, αλλά δεν υπάρχουν ουσιώδεις προοπτικές αλλαγής. Πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε σοβαρά την αναθεώρηση των πολιτών προοπτικών. Πρέπει να προπαρασκευαστούμε για αυτή τη μάχη που σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη και η άλλη μάχη που πρέπει να δώσουμε θα είναι η έκθεση για τις, ε, τους περίφημους ίδιους πόρους. Να δούμε κατά πόσον είναι πραγματικά ήδη οι πόροι ή πόροι των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πράγματι πρέπει να προετοιμάσουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση, το Midterm Review και θα το συζητήσουμε αυτό το Σεπτέμβριο, μετά τι διακοπέ. Ο κ. Φερνάνδε έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή απόψεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη, στεναρή υποστήριξη για να δώσει τη μάχη όταν επιστρέψουμε μετά τι διακοπέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν θα επιστρέψουμε λοιπόν, μετά τις διακοπές, τις θερινές, θα έχουμε ένα έγγραφο εργασίας που θα αφορά τη θέση του Συμβουλίου, θα είναι ένα πλήρες έγγραφο, το οποίο το προετοιμάζω με τη βοήθεια της Γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα έχετε λοιπόν, όταν ξαναρχίσουν οι εργασίες, ένα έγγραφο πληρέστερο. Αν δεν ξεκινήσουμε προγράμματα. και αν δεν ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί δεν θα υπάρξει εκτέλεση. Αν δεν υπάρξει εκτέλεση τότε τελικά ίσως να υπάρξει πρόταση για τη μείωση των προγραμμάτων γιατί θα υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τι γίνεται με την απορρόφηση προσεκτικά και μπορεί να πει κανείς ότι ορίζον 2020 δεν εκτελείται σωστά. Αν καθυστερήσουν οι διαγωνισμοί, η υποβολή προτάσεων κλπ, είναι προφανές ότι εν συνεχεία δεν θα υπάρχει και εκτέλεση σωστή των προγραμμάτων. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράμματα, στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας Φερρυπίν, από τα 76 προγράμματα μόνο 37 υιοθετήθηκαν. Είναι σαφές ότι αν δεν υιοθετήσουμε κανένα δεν θα υπάρξει καμία εκτέλεση στον τομέα της συνεργασίας της εδαφικής. Τα περίπου 500 προγράμματα παρουσιάστηκαν και τελικά οθετήθηκαν μόνο τα 368 από τα 500. Λοιπόν, Έχουμε βέβαια το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, από την περίοδο 2014 μέχρι 2020. Μπορούμε να μιλήσουμε την πολιτική συνοχή σε ένα πλαίσιο πολιτές 2007-2022. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα στις περικοπές της δημοσιονομικές, αναφέρθηκα στο κεφάλαιο 1β, σε πληρωμές έχουμε 120 εκατομμύρια ευρώ, υποχρεώσεις πληρωμών, και 43,5 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας. Είχαμε μειώσει όσον αφορά τα κονδύλια για την περίοδο 2007-2013. Μετά μιλήσαμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου 45,6 εκατομμύρια για τις πληρωμές. μετά για το πρόγραμμα LIFE έχουμε 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχουμε μειώσεις παραδείγματο χάρη για τα φρούτα και το γάλα για τα σχολεία ή τα μέτρα για τις ε, άμεσες πληρωμές. Για να απαντήσω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που μετέθησαν όσον αφορά τον προγραμματισμό των πληρωμών. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Ξεκινά από μια αρχή. Δηλαδή, έχει επιτευχθεί μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε περικοπές όσον αφορά τις πληρωμές που θα υπονόμευαν μία ε, συμφωνία. Ενώ έχουμε αποδεχτεί ότι στις πιστώσεις πληρωμών δεν υπάρχουν αυτά τα συμπληρωματικά 2 δις ευρώ. Τώρα για να έρθω τώρα στην, στην Ελλάδα και τα 35 δις ευρώ. Λοιπόν, το μόνο που ξέρουμε για την ώρα γι' αυτό είναι οι ανακοινώσει στον τύπο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν έχουμε καμία πληροφορία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον αντίκτυπο. Το 2016, παραδείγματος χάρη, Δεν ξέρουμε πώς θα μοιραστούν τα χρήματα, το ποσοστό της συγχρηματοδότησης, ε, εάν θα τροποποιηθεί ή όχι ο κανονισμός εκεί θα έχουμε 95% το πολύ. Λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε για περισσότερες πληροφορίες. Να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μετά θα υπάρχουν διάφορες λύσεις, διάφορες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάποια πρόταση, ούτω ώστε να γίνουν σεβαστά τα στοιχεία της συμφωνίας όσον αφορά τα 35 δις ευρώ. Δεν είναι τίποτα και καινοφανές, παρόλα αυτά είναι μια πρόοδος, μια πρόοδος για την Ελλάδα για, από κάποιους σε κάποιους πόρους που προβλεπόταν ε, από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ίσως θα έχουμε διαφορετικές απόψεις πολιτικές, αλλά έχουμε κοινό στόχο, δηλαδή το σεβασμό της εντολής που μας έχει ανατεθεί από την ε, Ολομέλεια. Όλοι υπερψήφισαν τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία υπερψήφισε, ε, όλα τα κοινοβούλια ε, στηρίζουν τους στόχους και νομίζω ότι εδώ δίνουμε ένα μεγάλο παράδειγμα δημοκρατίας ε, και σεβασμού ανηλυμένων υποχρεώσεων. Και σε αυτό το πνεύμα θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο να τηρήσει τις θεσμεύσεις στο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει τελικά να ταιριάζουν, να συμμορφωθούμε με αυτά που λέμε. Να τα εφαρμόσουμε στις πράξεις και ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών οι χώρε εκείνες που συστηματικά καταψηφίζουν τον προπολογισμό, ακόμα και αν πριν είχαν υιοθετήσει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, να στείλουν κάποιο μήνυμα αυτή την περίοδο, ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο θα δούμε ότι δεν είναι ευρωσκεπτικιστέ. Είναι χώρε που τελικά υπερασπίζονται και την Ευρώπη και τι ανηλυμένε υποχρεώσει. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Ε, σας εύχομαι καλή ανάπαυση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να έχετε την απαιτούμενη δύναμη στην επιστροφή σας για να πετύχουμε αυτά τα οποία έχουμε στο νου μας. Όπως λειτουργούν τώρα τα ευρωπαϊκά όργανα, δίδουν επιχειρήματα στους ευρωσκεπτικιστές για το τρίτο τμήμα. Ο κύριος Ντεπρέ. Για, ε, μιλήσαμε για το τρίτο τμήμα, τώρα για τα υπόλοιπα τμήματα θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Ντεπρέ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που ήμουν απόν. Ήμουν για ψηφοφορίες στην Επιτροπή Λίμπε. Συνάδελφοι, θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα τμήματα κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μία και τα υπόλοιπα όργανα από την άλλη στο κεφάλαιο άλλα όργανα σχετικά με το Κοινοβούλιο. Εγώ σε μία βίβλο πιστεύω, σε αυτήν την οποία ψήφισε η Ολομέλεια. Επί τη βάση αυτού του κειμένου θα μου επιτρέψετε να προτείνω, συνάδελφοι, τις προτάσεις για τις διαφορετικές θέσεις του προϋπολογισμού. Θέλω εδώ να προειδοποιήσω ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα είναι κρίσιμα στις συζητήσεις που θα έχουμε για τον προϋπολογισμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αφορά το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε ήδη. Κοιτάξτε, το, το θέσαμε αλλά πολύ σύντομα, λέει ο Πρόεδρος. <coughs> Μετά από τη συνάντηση του Τριγωνικού Διαλόγου προχθές, υφιστάμεθα πολύ ισχυρε πιέσεις και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή σχετικά με το σεβασμό του άρθρου 27 που υπεγράφει κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και συμφωνίας της συμφωνίας της πολιετούς δημοσιονομικής. Καθορίζει με διαφορετικούς στόχους για κάθε όργανο, αλλά κυρίως 5% μείωση προσωπικού μέχρι το 17%. Αυτό σημαίνει ε, περίπου 1% το χρόνο. Ε, μας το υπενθύμησαν αυτό έντονα και εγώ ε, επιχειρηματολόγησα αντίθετα με ε, ζωηρό τρόπο αλλά δεν πάει να έχει τεθεί το πρόβλημα. Νομίζω πρόεδρε ότι θα πρέπει να κάνετε ένα διάβημα από πλευράς μας προς τον Γενικό Γραμματέα. Το ψήφισμα που έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημείο 40 ζητάει ολομέλεια από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει στην, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια πλήρη ανάλυση των θέσεων του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του τρόπου με τον οποίο ο στόχος μείωσης κατά 5% έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, όπως και του τρόπου με τον οποίο θα συνεχιστεί εμπροθέσμως η διαδικασία αυτή στα πλαίσια του οργανογράμματος. Θα υπενθυμίσουμε στο Γενικό Γραμματέα ότι η Ολομέλεια έχει καταθέσει το συγκεκριμένο αίτημα και είναι σημαντικό για μας για να μπορέσουμε να επιχειρηματολογήσουμε σωστά. Πόσο μάλλον που οι πιέσει στο επίπεδο του προσωπικού είναι πολύ σημαντικές γιατί δημιουργήθηκε και μια νέα πολιτική ομάδα. Σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων που ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η δημιουργία αυτής της νέας πολιτικής ομάδας έχει συγκεκριμένες συνέπειες σε επίπεδο χρηματοδοτικό και σε επίπεδο προσωπικού. Εάν δεν κάνω λάθος, η δημιουργία αυτής της νέας πολιτικής ομάδας, δεν αναφέρομαι στο ποιόν αυτής της ομάδας, αλλά μία επιπλέον πολιτική ομάδα αυτού του μεγέθους έχει σαν συνέπεια ένα επιπλέον αίτημα 43 θέσεων υπαλλήλων είναι ένα άμεσο θέμα και πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα καλύψουμε αυτές τις 43 θέσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε 43 θέσεις επιπλέον για να τις δώσουμε στους φίλους της κυρίας Λεπέν. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν προσωπικό. Τώρα, για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου σας είπα ότι είχα να πω. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή, ελεγκτικό συνέδριο, ευρωπαϊκό δικαστήριο. Μια παρατήρηση τεχνικού επίπεδου να κάνω πρώτα. Είναι πολύ πιο εύκολο για τα υπόλοιπα όργανα να εργαστούμε επί τη βάση εγγράφων του Συμβουλίου και όχι της Επιτροπής γιατί το Συμβούλιο για κάθε ένα από τα άρθρα τα δημοσιονομικά λέει ποια είναι βάση, ποια είναι η μείωση και πώς καταλήγουμε στο νέο ποσό. Ενώ αντίθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπαίνει στον κόπο να το κάνει, πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς μόνοι μας και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Τι ποσοστό δηλαδή αποτελεί η πρόταση μείωση και για, τουλάχιστον για μια φορά να μου επιτρέψετε να συγχαρώ το Συμβούλιο για την ποιότητα των εγγράφων που μας στέλνει. Εδώ υπάρχει μια περίεργη ανομαλία και εδώ θα ήθελα την άποψη των συναδέλφων. Δηλαδή, ε, για το ελεγκτικό συνέδριο, το ποσό το οποίο ζητείται από το ίδιο το όργανο είναι χαμηλότερο από το ποσό το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να του δώσει. Για το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν ζητά το ίδιο μία αύξηση 1,46% των πιστώσεων. Η Επιτροπή προτείνει 1,94%. Φαίνεται ότι αυτό συνδέεται με το ότι θα πρέπει να πληρωθούν κάποιες ασφάλειες για τις συντάξεις τις οποίες δεν είχε λάβει υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, κάθε φορά που πρέπει άλλα όργανα να πληρώνουν κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ξεχάσουν ε, τους τόκους ούτε σε σχέση με το συνολικό ποσό ούτε σε σχέση με την προσαρμογή αυτή. Τώρα πέρα από την συγκεκριμένη ανομαλία, κάτι το οποίο εδώ χαρακτηρίζω ασύμβατο με τα τεκτενόμενα γενικά, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι και το Συμβουλίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβαν υπόψη πλήρω το σύνολο των συνεπειών που προήλθαν από την αύξηση του αριθμού ε, των δικαστών ε, τα επόμενα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προβλέπεται κάποια αύξηση των πιστώσεων, αλλά δεν αρκεί να έχουμε συνεργάτες και δικαστές, θα πρέπει και η ε, μηχανή να ακολουθεί, δηλαδή να μπορεί να συνοδεύει η διοίκηση του δικαστηρίου την εργασία των νέων δικαστών γιατί υποτίθεται ότι αυτοί έχουν σαν στόχο ακριβώς να καλύψουν τις καθυστερημένες υποθέσεις. Το Συμβούλιο λοιπόν και η Επιτροπή δεν λαμβάνουν υπόψη το ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι απαιτείται μια ενίσχυση των μεταφραστών, σαν παράδειγμα, για τα έγγραφα τα οποία θα δοθούν στους νέους δικαστές. Αν οι νέοι δικαστές δεν μπορούν να έχουν έγκαιρα και γρήγορα τα έγγραφα στην ε, γλώσσα τους και ξέρετε ότι εδώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε οποιονδήποτε για μεταφραστή γιατί μιλάμε για πολύ συγκεκριμένη ε, γλωσσική ε, προσπάθεια ε, νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη συνέπεια. Όταν μπούμε σε λεπτομέρειες, σε άλλη φάση θα πω ότι είμαι πιο κοντά στο αίτημα του οργάνου και όχι τόσο στην πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Δεν έχω τώρα χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις εξωτερικές υπηρεσίε τη μία μετά την άλλη, αλλά να πω το εξής γύρω από το Συμβούλιο και λιγότερο μάλλον για την Επιτροπή. Για το Συμβούλιο όμως είναι σεφές. Ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη το Συμβούλιο και ποτέ δεν παίρνει σοβαρά τα αιτήματα για συμπληρωματικές πιστώσεις που καταθέτουν τα διάφορα όργανα στον τομέα της ασφάλειας. Εμείς επιλέξαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας με τα απαιτούμενα δημοσιονομικά μέτρα. Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται δεκτό από το Συμβούλιο και επίσης και σε ένα μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή. Αν τυχόν λοιπόν μπορέσουμε να δούμε τη συνολική εικόνα και μπορούμε να διαρθρώσουμε τις περικοπές τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, αλλά και το Συμβούλιο, να πω το εξή. συνολικά. Λιγότεροι υπάλληλοι. Οι μειώσει αφορούν τον αριθμό των υπαλλήλων λιγότερες αποζημιώσεις, μικρότερη κινητικότητα, λιγότεροι εξοπλισμοί και λιγότερες πάνε στον τομέα της ενημέρωσης. Δηλαδή θα έχουμε λιγότερους υπαλλήλου, οι οποίοι δεν θα έχουν τα απαιτούμενα μέσα για να δουλέψουν και δεν θα μπορούν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους γιατί όλες οι πιστώσεις σχετικά με την δημοσιότητα που δίδεται στις εργασίες μας μειώνονται. Λοιπόν, θα τα εξετάσω αυτά ένα προς ένα για να δω τι σημαίνει και θα σας παρουσιάσω μια πλήρη έκθεση για κάθε ένα από τα όργανα. Ταυτόχρονα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Συμβούλιο υπάρχει ένα δωράκι το οποίο δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ε, καλό κυρίως προς την, την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω και ενώ σε όλα τα υπόλοιπα όργανα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει περικοπές, μικρότερες από το Συμβούλιο, αλλά παρόλα αυτά κάνει περικοπές και σε σχέση με την κινητικότητα και σε σχέση με τον εξοπλισμό και σε σχέση με τους υπαλλήλους, εξαιρούν και ιδίω σε επίπεδο διοικητικό την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και ο κύριος Φερνάντες το είδε αυτό και στο ε, τρίτο τμήμα του προϋπολογισμού για το οποίο είναι υπεύθυνο. Θα επανεξετάσω λοιπόν τις ανάγκες της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων με τα ίδια τα επιχειρήματα κριτικής που χρησιμοποιήσει η Επιτροπή εις βάρος όλων των υπολείπων οργάνων. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας, Πρόεδρε, ε, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Για αυτά που είπε για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, μα είναι ε, μια υπηρεσία που πρέπει να εφαρμόσει την τόσο σαφή εξωτερική μας πολιτική. Όλοι ξέρετε ότι έχουμε εξωτερική πολιτική αστεία τα έλεγα. Όσοι θα πάρουν το λόγο, παρακαλώ να είναι σύντομοι. Γιατί οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν σε 11.30. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τις συζητήσεις μας για την έκθεση του κυρίου Φερνάντες ε, κοίταζα τα νούμερα για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και όντως εξεπλάγει πρέπει να το πω διότι αν δούμε το εισόδημα, ε, τα έσοδα μας το 14 βλέπουμε με διαφορά 22 εκατομμυρίων δηλαδή το 2016 θα έχουμε ε, λιγότερα έσοδα από το 2014 να δούμε τα διάφορα κεφάλαια για παράδειγμα 2,7 από ενίκια το 14 έσοδα. Τώρα βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά δεν βλέπω να ε, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Δηλαδή θα αυξηθεί το εισόδημά μας ε, από τη μια μέρα στην άλλη κατά 22 εκατομμύρια. Τώρα οι δαπάνες. Εξετάζοντας τις δαπάνες βλέπω ότι συνολικά 50-60 δις παραπάνω δαπάνες προβλέπονται. Άρα συνολικά θα έχουμε το 2016 80 εκατομμύρια παραπάνω. Γιατί λοιπόν δεν τα δαπανούμε για να πληρώσουμε για τα κτίρια μας πιο γρήγορα. Τι διαδικασίες είναι αυτές ασχολούμαι με τον προπολογισμό εδώ και πολλά χρόνια, με θέματα προπολογισμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για πρώτη φορά βλέπω αυτή την πολύ περίεργη ε, προσέγγιση ενό προπολογισμού και δεν βλέπω και για ποιο λόγο. Για παράδειγμα, εξωτερικέ υπηρεσίε. 50 εκατομμύρια αύξηση σε σχέση με το 2014, χωρί να προβλέπετε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εστιατόρια. Επιδοτούμε τα εστιατόρια μα 4 εκατομμύρια το 2014 ε, το επιδοτούσαμε, τα επιδοτούσαμε με 4 εκατομμύρια και τώρα το 16 θα είναι 1,36 αυτή η επιδότηση. Για ποιο λόγο θα υπάρξει κάποια άλλη διαδικασία προκήρυξης για τα εστιατόρια μας. Θέλω εξηγήσει. Δεν είναι σωστός τρόπος ε, κατάρτισης ενός προπολογισμού. Κάτι άλλο που ανέφερε ο κύριος Ντεπρέ και συμφωνώ απόλυτα είναι ότι πρέπει κάθε χρόνο να μειώνεται το προσωπικό κατά 1% όλων των θεσμικών οργάνων. Και τι έγινε στο Κοινοβούλιο μεταξύ του 2013 και του 2015 δημιουργήσαμε 44 νέες θέσεις εργασίας. Και παράλληλα διάφορες υπηρεσίες μας δίνονται σε εξωτερικούς ε, παρόχους υπηρεσιών και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό και πόσους απασχολούν. Αντί να μειώσουμε λοιπόν το προσωπικό μας θα μπορούσαμε να, το αυξήσουμε και δεν ξέρουμε ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες μας. Όσοι είστε εδώ από το 2009 θα θυμάστε ότι τότε είχαμε κάνει έναν ε, έλεγχο για δύο ε, γενικές διευθύνσεις, ασφάλεια και ε, υποδομές. Ήταν εσωτερικός έλεγχος. Ο έλεγχος έγινε από 12 υπαλλήλους που έκαναν έκθεση απευθείας στον Γενικό Γραμματέα. Τώρα δεν θέλω να επιτεθώ στον Γενικό Γραμματέα. Καλά είναι όλα αυτά η εσωτερική έλεγχη, αλλά δεν είναι δυνατόν ε, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τα αριθμητικά στοιχεία να διαχειριστούμε τον προπολογισμό και το Κοινοβούλιο γενικότερα. Οπότε θα ήθελα να κοιτάξετε τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας, την DG Safe, και ίσως να ζητήσουμε εξωτερικό έλεγχο στην ΣΕΙΦ μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου για παράδειγμα. Έτσι θα βοηθούσαμε νομίζω το Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει τη διαχείριση αυτών των τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως σκοπεύω να απευθύνω μια επιστολή στο Γενικό Γραμματέα. Είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί. Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από την δυνατότητα ελέγχου των δαπανών, ιδίω στο Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω να θέλει κανείς ε, άλλο το λόγο. Αυτό είναι καλό γιατί ε, έχουμε την υποχρέωση να τελειώσουμε μέχρι τι 11.30 γιατί μέχρι τότε προβλέπεται η διερμηνία. Κύριε Ντεπρέ, ε, πορίσματα. Ντεπρέ, ναι βεβαίω, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο συνάδελφο ε, κύριο Μάνκα. όντω. ο γενικό γραμματέα πρέπει να παραστεί ενώπιόν μας και για το θέμα του προσωπικού και για τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Μάνκα για να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Ναι, μεν δεν υπήρξαν ε, άλλες παρεμβάσεις τώρα, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρξουν αργότερα. Ναι. Μπορούμε τώρα να εξετάσουμε το διορθωτικό προπολογισμό του 2015. Η κυρία Ζαμπάλ, αν έχει την καλοσύνη, θα μπορούσε να μας πει τι γίνεται με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού για το 2015. Eh, Η κατάσταση προς είναι ότι θα κατατεθεί ο έκτος διορθωτικός όπως σε όλα τα χρόνια είναι μια τεχνική διά, ε, διόρθωση των ιδίων πόρων ξέρετε ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε αυτή την πρόταση η οποία κάπως ε, θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να, να μειώσουν συγγνώμη, τις ε, συνιστής, ε, συνεισφορές τους κατά 892 εκατομμύρια ευρώ διότι υπάρχουν έσοδα κάπως μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ένας νέος, αν θα υπάρξει μια επιπλέον τέτοια διορθωτική επιστολή. Τα σχόλια που έχουμε είναι ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα και αυτό θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα το ύψος των συνεπειών που θα έχει κάτι τέτοιο και δεν έχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για να κατανοήσουμε αν κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τον παρόντα προϋπολογισμό. Υπάρχει επίσης η κινητοποίηση και ενός νέου ταμείου αλληλεγγύης, το οποίο καταρχάς, αν και δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, δεν θα είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε μια νέα διορθωτική επιστολή. Με τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη κινητοποιηθεί στο παρελθόν υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη αυτής της ε, διορθωτικής επιστολής. Αυτά θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο επιπλέον πρόβλημα. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, απλά διορθωτικό για τους ιδίους πόρους υπαριθμών 6. Σας ευχαριστώ για τις Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε μετά τις διακοπές. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα της Ελλάδας και τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν. Δεν ζητά κάποιος το λόγο όσον αφορά τη χρήση 2015, οπότε ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα όσον αφορά τον προπολογισμό. Ο κύριος Γενικός Εισηγητής τώρα ας μας ενημερώσει επί των πιλωτικών προγραμμάτων, επί των προπαρασκευαστικών δράσεων επίσης. Έχουμε έχουμε αύξηση των προτάσεων, κάτι που δείχνει το ζήλο των βουλευτών, τη φαντασία που δείχνουν, που έχουν, την βούλησή τους να ανοίξουν νέους δρόμους, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολιτών. 303 τήσεις υπερβλήθησαν, διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πέρσι. Χωσέ Μανουέλ, θα μπορούσατε να μας πείτε ε, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτό. Διότι αυτά τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να κατατεθούν υπό τη μορφή τροπολογιών του προπολογισμού και θα πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι, όσον αφορά το θέμα, πρέπει να ετοιμαστούν όλα αυτά μέχρι τη Σεπτεμβρίου και πιστεύω δέκατο του για τις πολιτικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ο αριθμός των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών ε, προγραμμάτων δείχνουν το ενδιαφέρον που έχουν οι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ίσως. Θα μιλήσω γαλλικά, λέει ο κύριος Συγητής. Έχουμε 303 προτάσεις λοιπόν. 269 πιλωτικά προγράμματα και 39 προπαρασκευαστικέ ε, δράσεις. Πράγματι, οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι τροπολογίες πολιτικές ομάδες μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κατατεθούν λοιπόν οι τροπολογίες μέχρι τότε. Έχουμε πολύ περιπλησμένα περιθώρια, το υπενθυμίζω. Λοιπόν, Υποχρησιμοποιούμε το μέσο ευελιξίας λόγω της από αποθεματικών και περιθώριων. 40 εκατομμύρια έχουμε σαν μέγιστη δυνατότητα για τα πιλωτικά προγράμματα και 50 εκατομμύρια για τις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις. Αυτά τα πιλωτικά σχέδια, αυτός ο κατάλογος φτάνει στα 339 εκατομμύρια αδύνατο να πετύχουμε το στόχο. Έχει γίνει μια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 30 προγράμματα, 19 πιλωτικά και 11 ευρωπαρασκευαστικές δράσεις. Δίνει τον καλύτερο βαθμό Α, 45 προγράμματα στη βαθμολογία Β, 173 σε και 43 με βαθμό D. και θα πρέπει να κάνουμε τη δέουσα εξέταση. Εγώ προτείνω και συστήνω να προσπαθήσουμε τα, τις ε, που έχουν τη βαθμολογία Β να προσπαθήσουμε να περάσουμε στο Α. Όλα τα προγράμματα είναι σημαντικά, μπορούν πάντα να βελτιωθούν, είναι σημαντικά όλα για να έχουμε καλύτερη ποιότητα, πιο συνολική προσέγγιση, καλύτερη ποιότητα στον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ανέφερθηκα στα αποθεματικά που είναι ελάχιστα. Επιμένω επί της υποβολής των τροπολογιών ε, όσον αφορά τον προπολογισμό στην κατηγορία 1α το Κοινοβούλιο έχει 86 πλωτικά προγράμματα και 11 προπαρασκευαστικές δράσεις 7 προγράμματα α 13 στο Β και 47 στο ΣΕ. Στην 1Β έχουμε 11 πολιτικά προγράμματα και 8 προβασιβαστικές δράσεις, 6α και ένα πρόγραμμα με το βαθμό Β. Στο κεφάλαιο 2 έχουμε 72 πιλωτικά προγράμματα, 3α, 13β, 51σε, κατηγορία 3, 67 πιλωτικά, 9 προπαρασκευαστικε δράσει, δράσεις 6α14β 41C και πάρα 4 το Κοινοβούλιο παρουσίασε 25 πιλωτικά προγράμματα 6 δράσει προπαρασκευαστικε 21C κατηγορία 5 έχουμε 3α 2β ψηλωτικά προγράμματα και ένα c κατηγορια 5 εχουμε 3 α 2 β ψηλωτικα προγραμματα και ενα ΣΕ. Έχουμε τους περιορισμούς που σας υπενθύμησα, δεν έχουμε διαθέσιμο αποθεματικό και περιθώριο. Βεβαίως θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε τα αναγκαία περιθώρια σε όλες τις κατηγορίες, τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Ήδη έχουμε την αξιολόγηση, θα βοηθήσει να κάνουμε την ε, επιλογή των διαφόρων ε, προγραμμάτων και γι' αυτό κάλεσα, ζήτησα τα προγράμματα που είναι στο Β να περάσουν στο Α, στη βαθμολογία Α Όσον αφορά τα κατατεθέντα προγράμματα, ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να παρουσιάσουν πιλωτικά προγράμματα που μπορούν όπως πάντα λέω να βελτιωθούν. Βεβαίως υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα τα οποία κατετέθησαν όπου ήδη εκεί προσπαθούν να καλύψουν προγράμματα που καλύπτουν τα πιλωτικά προγράμματα ήδη. Ευχαριστώ όμως για την πρωτοβουλία, ευχαριστώ για την ποιότητα των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων που κατετέθησαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ. Τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες εκεί όπου τα περιθώρια μας είναι κάπως μεγάλα. Και όπου δεν υπάρχουν περιθώρια να προσπαθήσουμε να τα βρούμε. Σχετικά με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά καλούνται τις επόμενες έξι εβδομάδες που μας χωρίζουν από τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι ίδιοι λοιπόν οι υπεύθυνοι θα πρέπει να καταθέσουν τροπολογίες για να διευκολύνουν το πέρασμα στην κατηγορία 1 αυτών που κατηγοριοποιούνται Β, Γ και Δ σήμερα. Αυτά για τα πιλωτικά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα στο οποίο να σταθούμε ε, και θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα για τα της Μεσογείου και για την ολιστική συνολική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών φαινομένων. Το λόγο έχει ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα παρουσιάσω το σύνολο της κατάστασης στη Μεσογείο, θα ήταν πολύ φιλόδοξο, αλλά θα καταθέσω μία γνωμοδότηση ε, προς την Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών μετά από την έγκριση από πλευράς της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για τα θέματα της μετανάστευσης. Η γνωμοδότηση την οποία προτείνω και η οποία σας έχει αποσταλεί περιλαμβάνει βασικά τρία βασικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός φιλοδόξου, σχετικά φιλοδόξου προγράμματος γιατί κάποιες πολύ σημαντικές υποθέσεις και πλευρές δεν λαμβάνονται υπόψη. Αλλά υπάρχει μια κάποια φιλοδοξία στον τομέα της επανεγκατάστασης και μετακίνησης. Ξέρετε ότι προβλέπονται 40.000 μετακινήσεις και 20.000 επανεγκαταστάσεις για τις ε, κατηγορίες αυτές. και αντίστοιχα προβλέπονται και τα συμπληρωματικά δημοσιονομικά κονδύλια. Λοιπόν, από το 5 και 6 της πρότασής μου ζητώ και εδώ θα ήθελα να με στηρίξετε. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια σωστότερη αξιολόγηση, γιατί τα πράγματα τα βλέπουμε βραχυπρόθεσμα. Η προοπτική μας είναι ένα έτος, αλλά δεν θα σταματήσει το φαινόμενο αυτό σε ένα χρόνο το Frontex μπορεί να κάνει κάποιες αξιολογήσεις για τις μεταναστευτικές ροές τα επόμενα χρόνια. Και μιας λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε και για το θέμα της αναθεώρησης των δημοσιονομικών πολιτών προοπτικών, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση των αναγκών οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν αύριο, ιδιαίτερα για το, για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Είναι σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε ε, να ε, καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Θέλω να αλλάξει και η ονοματολογία η οποία ε, αφορά το συγκεκριμένο κονδύλι. Βλέπει κανείς ότι η νομική βάση η οποία επιτρέπει τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις του ταμείου αυτού, του ταμείου ΤΑΜΕ όπως λέμε ελληνικά, ε, μεταφράζεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά τα οποία θα πρέπει ε, να χρηματοδοτηθούν αλλά δεν ανταποκρίνονται και δεν αντιστοιχούν στην κοινοτική ονοματολογία. Η κοινοτική ονοματολογία έχει παραμείνει σε ένα προηγούμενο στάδιο πριν τη δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου. Αυτό που θα μας επιτρέψει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και να ελέγξουμε καλύτερα τις πιστώσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε την ονοματολογία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε στο εσωτερικό του ταμείου τα διαφορετικά επιμέρους προγράμματα και τα δημοσιονομικά μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας όπως και την δημοσιονομική ευελιξία. Το τελευταίο τμήμα, και εδώ έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Γκέγερ, την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με ευφυή τρόπο τις εξωτερικές υπηρεσίες όπως την ΕΑΣΟ και το Frontex. Έτσι και αλλιώς η ΕΑΖΟ αντιμετωπίζεται με κάπως διαφορετικό τρόπο, αλλά τη Frontex, σαν παράδειγμα, τη μία χρονιά τους δίνουμε κάποιο προσωπικό επιπλέον και την επόμενη τους το παίρνουμε πίσω. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Και ακόμα και για ε, υπηρεσίες οι οποίες αναλαμβάνουν αποστολές ε, τις οποίες χαρακτηρίζουμε στρατηγικού ενδιαφέροντος. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Αυτές είναι οι ε, προτάσεις τις οποίες κάνω στην Επιτροπή και που θα κάνω στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Θα γίνει μια σύντομη συζήτηση. Ζάμπαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Δεπρέ στην παρουσίασή του για την γνωμοδότηση, είπε ότι ζητάει τη στήριξη της ε, Επιτροπής, συμφωνώ, η Σοσιαλιστική Ομάδα στηρίζει αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί συμμεριζόμεθα όλα τα σημεία που θέτει και ιδιαίτερα ότι θέλει να γίνει αυτή η αποτίμηση για το μέλλον, για να δούμε τι ανάγκες ε, θα έχουμε για να ενημερωνόμεθα καλύτερα και να έχουμε καλύτερα στοιχεία όταν θα υποβάλουμε την πρόταση αναθεώρησης των πολιτών προοπτικών. Έχετε τη στήριξη της ομάδας μου και θα υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεσόφσκι. Ο κύριος Δεσόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς ε, του ΕΛΚ και εμεί στηρίζουμε την πρόταση του κυρίου Ντεπρέ. Η αύξηση του προπολογισμού για την Frontex και το ε, ΕΑΣΟ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξη για το Άσυλο, είναι αναγκαία, αλλιώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση μετανάστευσης και πρέπει, όπως και η Europol και η Eurojust, να εξαιρεθεί από τη μείωση του προσωπικού. Στηρίζουμε λοιπόν και αυτή την πρόταση. Να μην υπάρξει μείωση προσωπικού. Και γενικότερα πρέπει να δούμε πώς τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι περικοπές προσωπικού γιατί αυτοί οι εξωτερικοί οργανισμοί έχουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να περικόπτουμε το προσωπικό τους. Και χθε το συζητήσαμε. Η Eurojust οπωσδήποτε, όπως ακούσαμε λοιπόν χθε, μας εξηγήθηκε ότι η Eurojust ε, έχει όλο και περισσότερες συνεδριάσει. Μας είπαν για παράδειγμα ότι οι συνεδριάσει που χρειάστηκαν να οργανώσουν φέτος μέχρι τούδε ε, είναι περισσότερες από όσες έκαναν πέρυσι συνολικά. Άρα χρειάζονται μεγαλύτερο προπολογισμό για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον τομέα της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω εδώ μια έκθεση του οργανισμού φαρμάκων. Μην υποτιμήσετε. Εγώ έχω εργαστεί στον τομέα αυτό Συγγνώμη, δεν είναι οργανισμό φαρμάκων, είναι οργανισμό για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Εγώ έχω εργαστεί ε, ω κοινωνικό λειτουργό στο δρόμο και διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι ιδίω νέοι παίρνουν ή δοκιμάζουν νέα συνθετικά ναρκωτικά. Και πολλέ ε, παράνομε ουσίες εμφανίζονται στου δρόμου των πόλεων μα. και πολλέ φορέ δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προκλήσει. Η εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά αυξάνεται και γίνεται όλο και χειρότερη. Πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε. Άρα θα ήθελα για τον οργανισμό αυτό να υπάρξει αύξηση του προπολογισμού του οργανισμού αυτού EMCCD για να καταπολεμήσουμε τα αρκωτικά, τις ψυχοτρόπες ε, και ψυχοενεργές ουσίες. Πρέπει λοιπόν να κάνω μια έκκληση στον κύριο Ντεπρέ να λάβει υπόψη αυτό το αίτημά μου και επίσης καλό και τους συναδέλφους μου από τους σοσιαλιστές και άλλες πολιτικές ομάδες παρακαλώ να υποστηρίξετε αυτήν την αύξηση του προπολογισμού του οργανισμού για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Διότι μέχρι το πρόσφατο παρελθόν είχαμε μια πτωτική τάση χρήσης ναρκωτικών, αλλά τώρα έχει αντιστραφεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί το έτοιμά σας. Φανά. Ευχαριστώ. Από πλευράς Πρασίνων και εγώ θέλω να υποστηρίξω κατηγορηματικά και να χαιρετήσω αυτήν την γνωμοδότηση. Συμφωνούμε με όλες τις, ε, όλες τις ρήτρες για το 7, για την Frontex. Θα κάνουμε μια τροπολογία. Πρόσφατα συζητήσαμε με τον επικεφαλής της ε, Frontex και χαιρετίζουμε την αύξηση των πόρων ε, της Frontex, αλλά ανησυχούμε για τα, αρμοδιο... για τα καθήκοντα της Frontex. Ο Διευθυντής ε, μας είπε ότι θέλει η πρώτη προτεραιότητα να είναι η διάσωση, αλλά στην εντολή της Frontex αναφέρεται η προστασία των συνόρων ως κύρια αρμοδιότητα. Αναφέρεται την εντολή στο 7, αλλά ασχολείται μόνο με την πολιτική επαναπροώθησης. Οπότε θα θέλαμε να κάνουμε μια τροπολογία για να είναι πιο ευρία η εντολή και συγκεκριμένες προτεραιότητες της Frontex. Υποστηρίζουμε αυτό που πάντα ζητούσαμε επίσης, το ότι πρέπει να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του, του γραφείου για το άσυλο. Λέτε κι εσείς ότι πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη, άρα πρέπει να έχει περισσότερους πόρους. Ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια κοινή πολιτική ασύλου. Πολύ σημαντικό είναι αυτό και γι' αυτό και αυτός ο φορέας πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης κρίσεων. Πρέπει όντω λοιπόν να λάβει περισσότερες πιστώσεις. Χαιρετίζω λοιπόν, ε, εκτός από αυτή τη μία τροπολογία, τη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ, κυρία Μυριάτα. Και εμεί θέλουμε να στηρίξουμε τα όσα είπε και ο Σντιπρέ. Είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση κατά την άποψή μου. Κάποια πράγματα θίξατε τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουμε. Η όλη αξιολόγηση είναι ένα και πώς οι υπηρεσίες συνεργάζονται μία με την άλλη, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει έλεγχος. Είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογηθεί, να ξοδεύονται και να σπαταλιώνται χρήματα άμα δεν ξέρει που πήγαιναν τα χρήματα. Πρέπει να πηγαίνουν στο σωστό σκοπό και θα ήθελα να ξέρω καλύτερα τα προγράμματα αυτά της ένταξης, περί τίνος πρόκειται, πόσο αποτελεσματικά θα είναι, ούτως ώστε να έχουμε μια μακρόπνοη θεώρηση των πραγμάτων για να πετύχουμε τους στόχου μας. Υποστηρίζω πλήρως λοιπόν ε, με αυτά που μας είπατε και με τη γνωμοδότηση σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ω Κολμέλο, τελευταίο που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο Ντουπρέ για αυτό το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Μία συμπλήρωση. Ο τίτλος λέει «Ενιαία προσέγγιση για την ε, κατάσταση στη Μεσόγειο. Μια ολιστική προσέγγιση. Ολιστική προσέγγιση σημαίνει ευρείες νέες δυνατότητες. Για παράδειγμα, έγκαιρα να βοηθούμε τους ε, πρόσφυγες και να τους ενημερώνουμε για να μην ξεκινάνε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε όμως ε, τις αναγκαίες πιστώσεις γιατί αλλιώ θα είναι απλώς ε, ευσεβής πόθη. Οπότε, στον τομέα αυτό, θα ήταν σκόπιμο, πιστεύω, να προβλέψουμε κάποιες πιστώσεις, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Γιατί οι διαπραγματεύσεις πάντα θα αφορούν χρήματα, διότι ε, δι χρημάτων. Εάν λοιπόν δεν έχουμε αποτέλεσμα με τη δράση μας και χάνουν τη ζωή τους αυτοί που επιχειρούν αυτό το ταξίδι, πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ θα μπορούσαμε ε, με πολύ καλό τρόπο να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις παρατηρήσεις κύριε Ντεπρέ για να ολοκληρώνουμε το θέμα. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους για τις εκτιμήσεις που εξέφρασαν, θετικές εκτιμήσεις σε αυτό το στάδιο. Θα εξετάσω όλες τις τροπολογίες με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό κείμενο, το οποίο να οδηγήσει στη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Λε Πρόεδρος. Τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν πριν τις 3 σήμερα το απόγευμα. Ως 3 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και ότι η Επιτροπή Λίμπε θα αποφανθεί πιθανότατα 16 Νοεμβρίου. Ερχόμαστε τώρα στις ψηφοφορίες και πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες θα ήθελα να κάνουμε μια δοκιμή, να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί το ηλεκτρονικό μας σύστημα ψηφοφοριών. Αν έχετε την καλοσύνη να βάλετε την κάρτα σας στην εισδοχή, στη συσκευή, θα κάνουμε μια πρώτη δοκιμή. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Μας λείπουν τέσσερις ψήφοι. 27 κάρτες έχουν εισαχθεί. 24 όμως ψήφους έχουμε. Τρεις από εσά ε, δεν έχετε πατήσει. Θα περιμένουμε. Δεν έχετε τις κάρτες σας. Έχετε την κάρτα σας. Θα προσθέσουμε λοιπόν την ψήφο σας. 25 λοιπόν είμαστε. Φτάσαμε. Κοιτάξτε. Ψηφίσατε όλοι. Εκείνοι που έβαλαν τις κάρτες τους. Ψήφισαν. Όχι. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Α, εντάξει, τα καταφέραμε. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Η πρώτη ψηφοφορία. Το σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης έκθεση της κυρίας Γκράσλε. Κυρία Γκράσλε, μια σύντομη σύνοψη πριν ψηφίσουμε, θέλετε, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Μονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Il un vote. Λείπει μία ψήφος. Κυρία Ντεπρέ, ψηφίζετε. Δεν λειτουργεί. Α, λειτουργεί, εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Προσθέτουμε μία ψήφο του κυρίου Ζανιέ. Λοιπόν, 27 ψήφοι υπέρ, μία αποχή, 28 ψήφισαν συνολικά. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Πάμε λοιπόν τώρα στο τμήμα 3 για το 2015. Κυρία Καδιαζαμπάλ, θέλετε να πείτε κάτι όσον αφορά τις προτάσεις ε, μεταφορών που έχουν προταθεί. Ευχαριστώ. Τρεις προτάσεις μεταφορών, 20, που έχει να κάνει με τη Συμφωνία Αλληλείας με τη Σενεγάλη, περίπου 11 εκατομμύρια, 24, κινητοποίηση της, ε, του αποθεματικού για την ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στη Συρία και τις γειτονικέ χώρες όπου ζητάμε 50 εκατομμύρια και 23 που την άφησα τελευταία γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο ε, ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση ε, ζητάμε να μεταφέρουμε 15 εκατομμύρια 15 εκατομμύρια και μισό διότι οι γραμμές του μέσου της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη έχουν ε, εξαντληθεί. Ζητάμε 15,5 για την επιστημιστική ασφάλεια με ημερομηνία 6 Ιουλίου. Για τις 6 Ιουλίου έχουν δαπανηθεί το 95% των πιστώσεων και για τη γραμμή για τους ε, μη κρατικού φορείς για την ανάπτυξη που έχει δαπανηθεί 186% και άλλο για το περιβάλλον και την διαχείριση των φυσικών πόρων όπου έχουμε δαπανίσει το 78%. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε το θέμα πληρωμών που έχουμε. φτάνουμε τώρα στη μέση του χρόνου και χρειαζόμαστε ήδη μεταφορές, γιατί η Κομισιόν δεν έχει πλέον πόρους για αυτές τις γραμμές. Ένα στοιχείο στην επιστημιστική ασφάλεια, όπου θέλουμε να βάλουμε 9,5 εκατομμύρια, η αρχική γραμμή είχε 140 εκατομμύρια. Και από αυτά τα 140, 45 χρειάστηκε για να πληρωθούν προηγούμενες ε, αποδείξεις. Παρακαλώ λοιπόν και για τις τρεις μεταφορές ε, για τη θετική σας ψήφο. Σας ευχαριστώ. Να ψηφίσουμε τις τρεις μεταφορές μαζί. Έχετε πρόβλημα. Δεν έχετε παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Κύριε Ζανή, Λοιπόν, 27 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Κυρία Ολμάιερ, Κυρία Ολμάιερ, για τους άλλα τμήματα θέλετε να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις που θα μας υποβάλλετε. Καταρχάς, η Γκρέσλε με ρώτησε και ο κύριος Κάιζερ, γιατί δεν έχω βέβαια όλα τα στοιχεία, στο καταστατικό των υπαλλήλων, κάποιοι λίγοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν προώρη συνταξιοδότηση για πολύ συγκεκριμένου λόγους. Είναι εδώ και ο Γενικό Διευθυντής Προσωπικού κ. Κάιζερ, μπορεί να μας τα πει, γιατί δεν ξέρω την ηλικία συγκεκριμένα. Εδώ μιλάμε για 9 άτομα και του χρόνου 7. Στην ουσία πρόκειται για δύο υπαλλήλου, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ 7 και 9, Οπότε πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες μεταφορές ε, πιστώσεων το κόστος είναι μικρότερο εάν, από το εάν έμεναν. Οι θέσεις αυτές δεν θα καλυφθούν μετά την αποχώρησή τους γιατί γίνεται μια αναδιάρθρωση υπηρεσιών γι' αυτό θα μειωθεί το κόστος ε, με τη συνταξιοδότησή τους δεν θέλω να αναφέρω ονόματα οπότε δεν είναι καταχρηστική αυτή η πρόταση, διότι καμία άλλη γενική διεύθυνση δεν ζήτησε να απασχολήσει τα άτομα αυτά. Νομίζω ότι ο κύριος Κάιζερ καταλαβαίνει τι εννοώ με αυτά που λέει και ελπίζω και εσείς να καταλαβαίνετε. προκύπτει δηλαδή ορισμένες φορές ότι ορισμένοι πάλι δεν χρειάζεται να μείνουν μέχρι το τέλος της καριέρας, του, καριέρας του. Γι' αυτό πρέπει να μεταφερθούν συγκεκριμένα ποσά την ηλικία των ε, ατόμων αυτών ε, δεν την ξέρουμε. Μήπως μπορείτε, μπορείτε να μας την πείτε. Ξέρω ότι μία κυρία εργαζόταν στην ομάδα ECR και το άλλο άτομο ήταν σε κάποια γενική διευθυνσή. Ο κύριος Κάιζερ μπορεί να μας τα πει. Γιατί αν πρέπει να αναφέρουμε ονόματα πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών γιατί δεν μπορούμε δημοσίως να αναφέρουμε ονόματα. Και είναι σωστό αυτό. Δεν θα ήταν σωστό να αναφερθούμε σε άτομα συγκεκριμένα σε δημόσια συνεδρίαση. Μήπως ο κύριος Κάιζερ μπορεί να μας εξηγήσει. Είναι 95.000 ευρώ που πρέπει να μεταφερθούν διότι ε, προκύπτουν ε, κάποιες δαπάνε από αυτήν την συνταξιοδότηση. Ο κύριος Κάιζερ. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο άτομο είναι 58 ετών. Από την 1η Ιουνίου έχει σταξιοδοτηθεί. Αυτό το μεταβατικό σύστημα ε, κράτησε 5 μήνες. Στην άλλη περίπτωση πρόκειται για έναν υπάλληλο που είναι 65 ετών. Ε, συγγνώμη, 56 ετών και θα αποχωρήσει οριστικά το Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για κάποιον που ασχολείται με την πληροφορική όπου επειδή χρησιμοποιούμε νέα συστήματα πληροφορικής δεν υπάρχει ανάγκη να παραμείνει στην υπηρεσία γιατί σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε να ενημερωθεί για τα νέα συστήματα πληροφορικής. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame vous estimez... Κυρία Χολμάιερ, εντάξει. Α, κυρία Αυτές τις ιστορίες τις παρακολουθώ για χρόνια, γιατί όταν ο συνήθις εργαζόμενο πρέπει να δουλέψει μέχρι τα 67 και εδώ οι υπάλληλοι μα φεύγουν 10 χρόνια νωρίτερα, αυτό είναι θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω σε τι βαθμό, σε τι βαθμό. Έτσι ξέρετε, για να έχω τα στοιχεία. Σε τι βαθμό είναι αυτοί που αποχωρούν. Ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού κ. Κάιζερ. Το βασικό, ο βασικός μισθός είναι AST, είναι κατηγορίες AST βοηθητικοί υπάλληλοι. Ο βασικός μισθός στη μία περίπτωση είναι 10.000 ευρώ και μειώθηκε στις 7.800 και μετά από δύο μήνες ε, στα 6.900 και το άτομο αυτό έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. Στην άλλη περίπτωση, σε αυτόν που είναι 56 ετών, για το άτομο που είναι 56 ετών, ο βασικός μισθός αρχικά ήταν 5.600, μειώθηκε λοιπόν μέσω τη χρήση αυτή τη δυνατότητα για του πρώτου τρει μήνε στα 4.700 ευρώ και μετά για του υπόλοιπου ε, τρεις μήνες στα 4.100 και τέλο στι 3.400. Η κυρία Φολμάια. Κοιτάξτε, κυρίως για την πληροφορική πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους ε, ποιους ε, προσλαμβάνουμε. Πρέπει να προσλαμβάνουμε άτομα που να μπορούν να εκπαιδευτούν. Να έχουμε άτομα που δεν μπορούν να εκπαιδευτούν σε νέες ε, τεχνικές, δεν έχει καμία έννοια. Όλα αυτά γίνονται με βάση τον δημοσιοπαλικό κώδικα και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο δεν μας προτείνει όπως πριν 7 άτομα παρά μόνο 2 γιατί αλλιώ και εγώ θα ενδιαφέρομαι να εργάζομαι έτσι να αποφύγουμε και μία επιμόλυνση του ΣΥΠΗΝ. Θα φροντίσουμε να είναι εξαιρετικές αυτές οι περιπτώσεις. Θα ήταν δημοσιονομικά επίφοβη μια μόλυνση του ΣΥΠΗΝ. Έχουμε διαφωτιστεί και πρέπει να τοποθετηθούμε για να επικυρώσουμε τη διάταξη αυτή. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε ονομαστική ψηφοφορία ποιοι είναι εκείνοι που είναι υπέρ, είναι υπέρ της έγκρισης αυτού. Ωραία, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και μία αποχή. Θέλετε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις τέσσερις ακόλουθες προτάσεις. Αφορούν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει ανάγκη ενίσχυση της ασφάλειας. Γι' αυτό χρειάζονται 150.000 ευρώ σε συγκεκριμένες σκάλες, είσοδο σε κάποιους χώρους, ε, χώρους ασφαλείας για να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Και υπάρχει και μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου να εισαγάγουν μια διαχείριση αποβλήτων, να υπάρχει καλύτερη επιλογή Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν και αυτές οι δαπάνες, 43.000 ευρώ, που θα προκύψουν από το 12.01 αμοιβέ και θα περάσουν σε μια γραμμή που αφορά τον εξοπλισμό των ε, αιθουσών και κτηρίων. 43.000 ευρώ λοιπόν πρέπει να μεταφερθούν από αυτή τη μία γραμμή στην άλλη. Αυτό είναι το πρώτο. Να τις πω όλες μαζί. Γιατί νομίζω ότι όλες είναι απλές. Να παρουσιάσω και τις τέσσερις αυτές μεταφορές. Ναι, ναι, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Επίσης, ε, χρειάστηκε να κάνουν περισσότερες ειδικέ εκθέσεις από ό,τι είχαν προγραμματίσει και μετά από δικά μας αιτήματα. Γι' αυτό χρειάστηκαν εξωτερικοί μεταφραστές, περισσότερες λοιπόν δαπάνες για γλωσσικά μαθήματα, που πρέπει να γίνουν, αυτό το επόμενο δηλαδή, και επίσης για τις υπηρεσίες καθαρισμού και ανακαίνησης, όλα όσα έχουν να κάνουν με τη συντήρηση επίσης, πρέπει να περάσουν σε ένα συμβόλαιο τύπου Omnium, δηλαδή όπως και στο Κοινοβούλιο μία υπηρεσία να τα κάνει όλα και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον 40.000 ευρώ. Συνολικά είναι 100.000 ευρώ όλα αυτά. 30.000 για το πρώτο σημείο, 30 για το δεύτερο και 40 για το τρίτο. Για τα εστιατόρια και τις καντίνες. Και μετά υπάρχει ένα άλλο σημείο για την επίσημη εφημερίδα πρέπει να αποσυρθούν 150.000 ευρώ και χρειάζεται πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί η επίπλωση γραφεία και καρέκλες για να ε, διατηρείται καλύτερη υγεία των υπαλλήλων 40.000 εδώ και επίσης θέλουμε να περάσουν από 4 σε 10 οι κοινόχρηστοι χώροι στο CAD 3 και εκεί χρειαζόμαστε εξοπλισμό, οθόνες και πίνακες για παρουσιάσεις. Δεν θα είναι λοιπόν μόνο σε αίθουσες συνεδριάσεων αυτές αυτός ο εξοπλισμός. Θέλουμε να μπορούν να συναντιόνται και σε άλλες, να γίνονται συνεδριάσεις και σε άλλες αίθουσες και χρειάζονται 30.000 λοιπόν ευρώ για να υπάρξει περισσότερο τέτοιος τεχνικός εξοπλισμός γιατί σε αυτές τις νέες τους νέους του χώρους για συνεδριάσει δεν υπάρχει αυτός, δεν είχε προβλεφθεί αυτός ο εξοπλισμός. Και επίση ε, στο 2114 συντήρηση και επιδιόρθωση των τεχνικών εγκαταστάσεων χρειάζονται περισσότερες δαπάνες γιατί εφόσον θα χρησιμοποιούνται τα, οι χώροι περισσότερο διότι έγινε μια ε, πλήρης ε, αναδιάρθρωση των χώρων συνεδρίασης χρειάζονται άλλες 15.000. Συνολικά λοιπόν 35.000. Και 5.000 ευρώ για καύσιμα γιατί χρειάστηκαν περισσότερα για μετακινήσεις με αυτοκίνητα και για την αγορά των αυτοκόλλητων για διόδια και 40.000 ευρώ για συμβούλους και ελέγχους για συγκεκριμένους επιμέρους τομείς. Αυτό είναι το τρίτο σημείο και άλλο ένα τελευταίο καθαρισμός και συντήρηση από εκεί παίρνουμε 110.000 και θα αξιοποιηθούν για να ενισχυθεί η ασφάλεια των κτίριων. Αυτό έχει να κάνει με το πρώτο σημείο το οποίο σας παρουσίασα στην πρώτη μεταφορά αλλά εδώ η μεταφορά γίνεται από άλλο σημείο του προπολογισμού, όπως σας είπα, από τον καθαρισμό και συντήρηση. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά 110.000. Αυτά ήταν όλα. Αν έχετε ερωτήσεις παρακαλώ, ακούω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Έγιναν τέσσερις, ε, τέσσερις ε, μεταφορές για τις πιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Παρακαλώ μπορούμε να ψηφίσουμε ο μπλοκ και για τα τέσσερα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Σκοτάει κλού. Πέρα ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Εξετάσαμε τις μεταφορές Έχουμε αιτήματα για μεταφορές από την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, δύο μεταφορές, κυρία Ελμάιερ. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα αυτό, μισό λεπτό για να βρω το έγγραφο. Α, πρόκειται λοιπόν για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ζητήθηκε μεταφορά επίσημη εφημερίδα. Α. Συγγνώμη για την Επιτροπή των Περιφερειών, λέει ο Πρόεδρος, σας ζήτησα πριν από την ΕΟΚΕ. Μισό λεπτό να το ψάξω να το βρω. Ψάχνω να βρω το, την Επιτροπή των Περιφερειών. Α, ωραία, σας ευχαριστώ. Επιτροπή των Περιφερειών πράγματι. Λοιπόν, 35.000 από προσωπικό και υπαλλήλου πάνε στις άδες, άλλες δαπάνες σχετικές με άτομα. 35.000 ευρώ λοιπόν. Διότι υπήρχε πλεόνασμα προσωπικού σε έναν τομέα και έλλειψη σε άλλο τομέα, οπότε γίνει και αυτή η μεταφορά. Προσπαθώ να βρω τα σχέδια δραστηριοτήτων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ τα έχω. Eine Sekunde. Das ist das Kicklass, oder? Χωρίς μικρόφωνο. Ich weiß nicht, wo das hier gelandet ist. Wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Χωρίτε, μπορείτε να περιμένετε λίγο. J'indique à ceux d'entre nous qui... Όσοι λοιπόν εξημών ε, θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα στην αντιπροσωπεία για τη Σικελία ...475.000 βοήθεια και συντήρηση των συστημάτων λογισμικού είναι η Επιτροπή Περιφερειών. Με συγχωρείτε που δεν τα ήξερα απ' έξω. Θέλουν ένα νέο σύστημα πληροφορικής να εισαγάγουν το οποίο είναι ασύμβατο και πολύ διαφορετικό με τα υπόλοιπα. Λέγεται κύκλος αυτό το σύστημα και θα αντικαταστήσει όλα τα ασύμβατα συστήματα ούτως ώστε να έχουν προς τα έξω και εντός ε, ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα για να δουλέψουν καλύτερα. Είναι 470.000 ευρώ που χρειάζονται λοιπόν και που θα λάβουν από άλλα σημεία του προπολογισμού τους και μας τα στέλνουν όλα αυτά μόνο για ενημέρωση. Τα θυμάμαι απ' έξω. Ε, γιατί το είχα συζητήσει αλλά δεν βλέπω το έγγραφο εδώ. Σας τα λέω απ' έξω. Και μια δεύτερη μεταφορά. Ναι, λέει η κυρία Χολμάε Το δεύτερο είναι μια μεταφορά που την ανέφερα. 35.000 για προσωπικό για να καλύψουν ε, τις ημερήσεις αποζημιώσεις και άλλες δαπάνες αποστολές λοιπόν είναι δαπάνες ε, για αποστολές 35.000 που θα πρέπει να μεταφερθούν από το κεφάλαιο υπάλληλοι και έκτακτοι υπάλληλοι. Από εκεί παίρνουν 35.000 και πάνε στις άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις δαπάνες των εργαζομένων στο θεσμικό ρένο 35.000. Εστώ εγκρίνεται τις δύο μεταφορές, μάλιστα. Ας ψηφίσουμε και τις δύο μεταφορές. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Και τώρα πρόταση μεταφοράς της ΕΟ και της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι, την είπα και προηγουμένως. Θα πάνε από την επίσημη εφημερίδα 65.000 για μελέτες, ακροάσεις και έρευνα. Για να κάνουν λοιπόν τέτοιες μελέτες και έρευνα χρειάζεται για να καλυφθούν τρεις μελέτες για τους εργαζόμενους και δύο μελέτες για την Συμβουλευτική Επιτροπή για βιομηχανικές αλλαγές για να υπάρξει η επιστημονική βάση για την ε, πολιτική τοποθέτηση. Δεν αυξάνονται λοιπόν τα, οι δαπάνες τους, απλώς γίνεται μια μεταφορά πιστώσεων. Δεν ζητά κάποιος το λόγο, οπότε θετική η σύστασή σας. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. το όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ και 3 ψήφοι εναντίον. Ενώ λοιπόν ετοιμάζεται την παρέμβαση σας κύριε αλμαίρ για την πολιτική της κληρονομιάς Λοιπόν, έχουμε τροποποίησει το προγράμματος, είχε γίνει ε, για την αποστολή στη Σικελία, οπότε μετά τη συνεδρίαση επιτροπής, όσοι θα συμμετάσχετε στην αποστολή, παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα. Κυρία Ολμάιερ, να μου κάνεις παρουσίαση. Δύο κτίρια. Α, για τα κτίρια. Λοιπόν, για τα κτίρια. Κάνε μια μεταφορά 7 εκατομμυρίων στον τομέα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει τον αναλυτικό κατάλογο του κόστους για τη διαχείριση των εργασιών για προσωρινές εγκαταστάσεις, υλικό, καθαρισμός, εξοπλισμός 92.500 για ορισμένες αλλαγές, για να εισαγάγουμε ορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό, δηλαδή τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας 570.000 και επίσης δαπάνες για να απομακρύνουμε τις παλιές εγκαταστάσεις και να αγοράσουμε νέες εγκαταστάσεις ασφάλειας πώς τα λέμε ακριβώς, αυτές οι θωρακισμένες ε, πόρτες, αυτό το γυαλί που είναι αλεξίσφαιρο, γιατί είδαμε επίσης ότι σε ένα επεισόδιο τραυματίστηκαν οι πάλι ασφαλείας, θέλουμε νέες πόρτες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να τις παραβιάσει, αλλά θέλουμε να είναι ε, διαφανείς αυτές οι πόρτες, να μην φαίνεται ότι έχουμε ταμπουρωθεί, να δείξουμε ότι είμαστε διαφανείς και φιλικοί προς τον πολίτη, αλλά ότι σεβόμαστε και την, ασφαλεία, την ασφάλεια συγγνώμη, του προσωπικού μας να μην μπορούν να τους ποδοπατήσουν. Ξέρετε τι έγινε, 300 Κούρδοι διαδηλωτές ορμήσανε, περάσαν τις πόρτες και δεν μπορούσε το προσωπικό μας να τους σταματήσει γιατί ήταν η φυσική πίεση τόσο πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και κοιτάξτε βέβαια, τίθεται και θέμα αξιοπρέπεια και γι' αυτό το Προεδρείο πήρε την απόφαση να ληφθούν όλα αυτά, να συνεχίσουμε να είμαστε διαφανείς αλλά και ασφαλείς, ασφαλέστεροι. Επίσης 530.000 γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια σε αυτά τα σημεία και επίση τον εξαερισμό, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν και επίσης και κατάλληλη υποδομή πληροφορική. και για να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε να αλλάξουμε κάποιους τείχους και ορισμένου εξοπλισμού 940.000. Όλα λοιπόν είναι 7,61 εκατομμύρια, 7,61 Μπορείτε λοιπόν όλοι να δείτε αναλυτικά ε, τι αποφάσισε το Προεδρείο και εμείς απλώς πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Διότι έχει ήδη γίνει μεταφορά. Έχει γίνει, έχει γίνει μεταφορά λοιπόν. Είναι μια επιβεβαίωση λόγω των ε, προβλημάτων ασφαλείας. Μια ερώτηση. Γιατί δεν τα είπαμε πριν τη συνεδρίαση. Για την κατανομή του κόστους. Εδώ βλέπω επιπλέον ένα εκατομμύριο για εργασίες που γίνονται εκτός των ε, συνήθων ωραρίων εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, ναι, και εγώ έκανα το ερώτημα αυτό. Μου είπαν, λέει η κυρία Χολμάερ, μου είπαν ότι πρέπει να εργαστούν. Α, παρακαλώ, μπορείτε εσείς, μπορείτε εσείς να με εξηγήσετε. Μήπως μπορεί η Γενική Διεύθυνση Υποδομών να μας πει, υποδομών και επιμελητίας να μας πει ο κύριος Έλιο Καρότσα. το 1 εκατομμύριο που προβλέπετε ήταν κάποιες επισκευές, κάποιες εργασίες πάρα πολύ στην είσοδο, ε, μόνο νύχτα, Σαββατοκύριακο και κατά τη διάρκεια των ημερών αδείας. Ε, γίνονται εργασίες εκτός ωραρίου εργασίας και αυτό κοστίζει επιπλέον λόγω των αμοιβών των εργατών. Αυτό το επιβάλλουν οι συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζομένους στο Βέλγιο. Όλμα, ε, ναι, μήπως μπορούσαν να γίνουν τον Αύγουστο, είπαμε, όπου δεν είναι κανείς παρόν. Μου είπαν όμως ότι δεν γίνεται, με το, για, λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το συμβόλιο. les travaux ne pas faire en août parce qu'on est en, Δεν μπορεί να γίνει τον Αύγουστο οι εργασίες γιατί είμαστε τώρα στα πλαίσια της ε, υποβολής εκδήλωση ενδιαφερόντων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβόλαιο για τη μελέτη της ε, συνολικής εγκατάστασης τα τμήματα των θυρών απαιτείται 10 με 11 εβδομάδες, οπότε το φινόπορο θα τα εγκαταστήσουμε. Πολ Μάια, θα πρότεινα, γιατί αυτό που λέει η κυρία Χόφμαν είναι όντως αιτιολογημένο, θα πρότεινα όταν βλέπω συνολικό κόστος ε, υλικού και εργασιών 6 εκατομμύρια και άλλο ένα από πάνω εκατομμύριο, πολύ ψηλό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το ένα εκατομμύριο να τονίσουμε ότι το αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα επικριτικά γιατί το σύνηθες κόστος εργασίας συμπεριλαμβάνεται στο άλλο ποσό. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο υψηλό το επιπλέον κόστος εργασίας, 60, συγγνώμη, ναι, 60% παραπάνω. Γι' αυτό θα πρότεινα ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να αναφέρουμε ότι οι εργασίες που θα γίνουν στις εισόδους πρέπει να γίνουν σε περιόδους που δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς επιπλέον και ότι το επιπλέον αυτό πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο διότι οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε περιόδους κατά τις οποίες αμείβονται κανονικά οι εργάτες. Κοιτάξτε, μπορεί να κουνάτε το κεφάλι σας, αλλά θα το αποφασίσουμε παρόλα αυτά. Δεν ξέρω αν είστε κατά τουλάχιστον ε, αυτό το αίτημα να μειωθεί αυτό το ένα εκατομμύριο νομίζω ότι έχει έννοια. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι στην ουσία παρακολουθούμε την επεξεργασία των θέσεων στις οποίες θα καταλήξουμε για να μειώσουμε το ποσό αυτής της σύμβασης. Ο κύριος Δεπρέ. Επί αυτού του τελευταίου σημείου, όταν εργάζεται κανείς στο Βέλγιο και εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι καταγεγραμμένες στο Βέλγιο, ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις. Και γενικά στο Βέλγιο γίνεται καλή δουλειά, ποιοτική δουλειά. Αν ο κόσμος εργάζεται το Σαββατοκύριακο, τότε οι αμοιβέ ορίζονται με διαφορετικό τρόπο. Αν τυχόν όμως εσείς εργάζεστε με αποσπασμένους εργαζομένους από άλλες χώρες, αυτό θα σας κοστίσει λιγότερο. Αλλά εφόσον θέλετε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες που διέπουν τις συλλογικέ συμβάσεις, τότε θα μου επιτρέψετε να θέσω το εξής ερώτημα. Διάβασα το σημείωμα, αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε ότι είναι απαραίτητο να κλείσουν και οι δύο βασικές είσοδοι ταυτόχρονα από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Τι θα γίνει, θα σκαρφαλώνουμε από τα παράθυρα, θα βάλετε εξωτερικές κλίμακες. Γιατί θα είναι απαραίτητο, λέτε, να κλείσουν ταυτόχρονα οι δύο βασικές είσοδοι. Βίρτς και Βάιλ. Ε, λοιπόν, από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Τι γίνεται, τεχνική άδεια, ε, έχετε κάνει λάθος, προβλέπετε κάποια άλλη λύση. Ο κύριος Καρότσα προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείσει φυσικά ε, το σημείο εισόδου. Γενικά, είναι μια γενική παρατήρηση. Εμείς θα επιταχύνουμε και ε, για να ε, μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα γιατί καταλαβαίνετε το να κλείσουμε την είσοδο αυτό θα κάνει τη ζωή δύσκολη όλων. Θα το κάνουμε αυτό ε, με περιόδους, ε, διακοπές. Θα το ρυθμίσουμε αυτό από τη Δευτέρα του Στρασβούργου μέχρι ε, την επιστροφή από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές από τις 7 λοιπόν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Ε, βλέπουμε λοιπόν να βλέπουμε ότι επελέγει η περίοδος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα γιατί από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει η Ολομέλεια μετά έχουμε διακοπές για τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά ακολουθεί η Πράσινη Εβδομάδα. Είναι ένας κοντός μήνας, τρεις εβδομάδες και θα κλείσουμε ταυτόχρονα λοιπόν και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σμικρύνουμε τη διάρκεια των εργασιών ενώ κανονικά θα χρειαζόμασταν μέχρι και έξι μήνες. Επιλέξαμε την περίοδο αυτήν στην οποία η κοινοβουλευτική δραστηριότητα δεν είναι ε, στις Βιξέλλες ή στο Στρασβούργο ή στις διακοπές. Κοιτάξτε, κάποιοι εργάζονται, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα μπαίνουμε στο κτίριο. Κύριε Ντεπρέ, ξέχασα να σας πω ότι προφανώς θα πάρουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε η κοινοβουλευτική δραστηριότητα να γίνει αντικείμενο εγγύησης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Είδατε ήδη διάφορες αφήσεις της εισόδους, ανακοινώνεται ότι θα γίνουν εργασίες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια λεπτομερής ανακοίνωση και για τα μέλη και για το προσωπικό έτσι ώστε να δώσουμε σε όλους την δυνατότητα να συνεχιστεί η κοινοβουλευτική δραστηριότητα χωρίς πολλά προβλήματα. Ε, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, κυρία Γκρέσλε. Μα πολύ περίεργο. Το καλοκαίρι που έχουμε 4-5 εβδομάδες όπου είναι πολύ μειωμένη δραστηριότητα δεν κάνατε έτσι την προκήρυξη που να μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την περίοδο. Να μου το εξηγήσετε αυτό. Χωρίς αυτή την τεράστια αύξηση του κόστους. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη μεταφορά. Εγώ δεν θα την είχα ψηφίσει. Μα μου είπατε ότι έχει ήδη γίνει η μεταφορά. Και εμείς απλώς πρέπει να την επικυρώσουμε για λόγους ε, δημοσιονομικής τεχνικής. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που κάνετε, έτσι να δαπανάμε χρήματα. Θα ήθελα να μας πείτε τι κάνετε για να μειώσετε περαιτέρω το κόστος σε σχέση με αυτό το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει η εναλλακτική λύση που πρότεινε η κυρία Χολμάιερ. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια είναι για, τα, για τον κάρτο των αχρήστων. Χολμάιερ. Να μην ξεχνάμε τι κάνουμε. Ε, εγκρίναμε μέχρι στιγμής μόνο 7 εκατομμύρια αυτή είναι απόφαση εντός του προπολογισμού, όχι για περαιτέρω δαπάνες. Και πιστεύω ότι στην απόφαση, μετά την πρόταση της συναδέλφου Χόφμαν, με την οποία συμφωνώ, και γιατί συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι αυτό το κόστος του επιπλέον ενός εκατομμυρίου μπορούμε να το μειώσουμε, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, αλλά είχα πει ότι πρόκειται να διορθωθούν τα σανσέρ μέχρι τον Αύγουστο. Και το κάναμε σε μια περίοδο που τα χρειαζόμασταν όλοι τα σανσέρ. Πιστεύω με την κυρία Γκρέσλε ότι θα ήταν δυνατόν να γίνουν οι συντηρήσεις των ασανσέρ τον Αύγουστο. Αλλά μας είπατε ότι τον Αύγουστο οι εργάτες έχουν διακοπές. Αλλά και εμείς κάνουμε διακοπές. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν μια κάποια ε, έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ε, διοίκηση του σώματος. Παρακαλώ και να μπει και στα πρακτικά ότι αυτό το επιπλέον κόστος ενός εκατομμυρίου πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Και οι εργασίες πρέπει να γίνονται όταν είμαστε στο Στρασβούργο. Τότε δεν χρειάζεται να εργάζονται νύχτα. Μπορούν να εργαστούν στις δύο εισόδους. Και οι, εργάτες να μπαίνουν, οι εργαζόμενοι να μπαίνουν από αλλού. Καταλάβαμε. Θα πρέπει στην επιστολή που θα στείλω στο Γενικό Γραμματέα πέρα από αυτά που εξέφρασε ο κύριος εισηγητής του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, θα προσθέσω και μια ιδιαίτερη αναφορά, δηλαδή στο μέγιστο δυνατό να μειωθεί το συμπληρωματικό κόστος. Κυρία Χόφμαν. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, να τελειώνουμε. Ναι, συμφωνώ με την κυρία Χόλμαν. Και αυτό ο κύριος Δεπρέ επίσης έχει δίκιο. Δεν θέλουμε να αφιζητήσουμε αυτό το 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως και η κυρία Χολμαέρ λέω, είναι υψηλό επιπλέον κόστος. Υπερβολικά υψηλό κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τις συλλογικέ συμβάσεις στο Βέλγιο. Αλλά όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, το θέμα είναι εάν αξιοποιούμε τους πόρους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοιτάξτε, θα το ρυθμίσουμε σήμερα, θα το παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγες. Η κυρία έθεσε ένα ερώτημα, δεν δόθηκε η απάντηση. Κύριε Καρότσα, θέλετε να απαντήσετε στις παρατήσεις της κυρίας ε, Γκρέστολ. Ψηφίσαμε τις πιστώσεις πριν έχουμε τις λεπτομέρειες ε, του όλου εγχειρήματο. Ίσως ε, δεν είναι η σωστή προσεγγίση. Λοιπόν, δεν έγινε δεν μπορούσε να διοργανωθεί η εργασία, ο διαγωνισμός οργανωθεί να γίνουν εργασίες τον Αύγουστο. Μαζί με τη Γενική Διεύθυνση ΛΟ και τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας χρησιμοποιήσαμε τα κατάλληλα μέσα του δημοσιονομικού κανονισμού που επιτρέπουν την κατεπίγουσα δικασία και παρά την κατεπίγουσα δικασία πρέπει να σεβαστούμε τις προθεσμίες του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εργασίες δεν είναι απλές, είναι σημαντικές, είναι μεγάλες οι δουλειές που πρέπει να κάνουμε και πιστεύω ότι η κυρία Ολμάγερ εξήγησε πολύ καλά ότι πρέπει να γίνουν οι εργασίες αλλά πρέπει να φαίνεται ότι επικρατεί διαφάνεια στο θεσμικό μας όργανο και χρειάζεται να είναι περίπλοκες οι εργασίες για να έχουμε και ασφάλεια και να επικρατεί και διαφάνεια. Κάναμε τα πάντα εδώ και μερικούς μήνες και πιστεύω χτες ή προχθές η Γενική Διεύθυνση Υποδομών έλαβε τις προσφορές από τρεις εταιρείες Λοιπόν, όλα γίνονται τόσο ώστε αυτού του μηνός να υπογραφούν οι συμβάσεις με μία από τις εταιρείε. Καλώς, είμαστε θύματα, κατά κάποιο τρόπο λέει ο Πρόεδρος, βασιλεύουν οι κανόνες, είμαστε το βασίλειο των κανόνων και κάποια φορά πέφτουμε θύματα των κανόνων μας. Είναι ο κανόνας των κανόνων. Λοιπόν, είναι ο κίνδυνος που δημιουργεί η γραφειοκρατία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι πιο φθηνές εργασίες και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ολοκληρωθεί η συζήτηση σε τρία λεπτά. Δεν θα έχουμε πλέον διαρμηνία, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρόταση. Διάρση τη χειρό. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά, λέει ο Πρόεδρος, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος ενάντιον και τέσσερις αποχές. Τελευταίο θέμα, κυρία Χολμάιερ. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ταϊλάνδη. Υπάρχει μια αλλαγή για την Ταϊλάνδη για τους εξής λόγους. Μειώθηκε το προσωπικό στην Ταϊλάνδη. Έχουν 30% λιγότερο προσωπικό. Το κτίριο έχει χρησιμοποιηθεί για 26 χρόνια και είναι πεπαλαιωμένα. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν το ανακαίνισε και στην ουσία θέλει να το κατεδαφίσει. Και η ασφάλεια στην περιοχή γύρω από το κτίριο έχει επιδεινωθεί και συνεργαζόμεθα με Συνεργαζόμεθα και με την ανθρωπιστική βοήθεια για να νοικιάσουμε ένα νέο κτίριο. Βρήκαμε ένα νέο κτίριο, δύο όροφοι σε ένα ε, κτίριο 34 ορόφων. Ε, είναι ο ένατος και ο δέκατος. Αντίθετα με το προηγούμενο, οι δύο όροφοι έχουν εσωτερική σκάλα που τη συνδέει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βγουν από το κτίριο οι πάλι όπως προηγουμένως και οι τουαλέτε επίσης, αντίθετα με ό,τι στο προηγούμενο κτίριο, είναι εντό του κτίριου. Γιατί ξέρετε, είναι δυσάρεστο να πρέπει να βγει κάποιο. Να χρειάζεται να βγει για να πάει στην τουαλέτα. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις νομίζω ότι καθιστούν σαφές ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτές οι δύο, τα δύο στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε κτίριο έχουμε 56 συνεργάτες άρα σεβόμεθα αυτά που χρειάζονται για τετραγωνικά μέτρα ανά ε, συνεργάτη. Επίσης ε, θα χρειαστούν 1,7 εκατομμύρια για εργασίες τα οποία θα περάσουν μετά στο νίκη. Το ενίκιο λοιπόν συνολικά για τα επόμενα 15 χρόνια θα είναι 14,4. Είπα λοιπόν ότι οι εργασίες θα κρατήσουν 3 χρόνια, θα κοστίσουν 1,7 εκατομμύρια και θα κάνουμε μια προχρηματοδότηση και το κόστος για ε, ίδρυυση, ηλεκτρισμό κτλ. είναι 2,8 άρα συνολικά 19,18 22 ευρώ τετραγωνικό μέτρο είναι χαμηλότερο από το μέσο κόστος το νίκη λοιπόν και το κόστος ε, για το ενίκιο συνολικά του κτηρίου δεν είναι υψηλότερο ενώ είναι πολύ καλύτερο το κτίριο. Η ΕΚΟ θα αναλάβει 25% της ενοικίασης και των λογαριασμών 4,7 εκατομμύρια λοιπόν θα πληρώσει η ΕΚΟ από το συνολικό αυτό κόστος οπότε νομίζω ότι είναι ε, πολύ καλός αυτός ο διακανονισμός Υπάρχουν ερωτήσεις δεν νομίζω ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, μία αποχή. Ολοκληρώσαμε. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Να σε ευχαριστήσω συνάδελφοι για το επιτελεστέν έργο. Το έργο που επιτελέσαμε αυτή τη χρονιά, σημαντική δουλειά. Σας εύχομαι θερμά έξοχες διακόπες. Λοιπόν, αν σας αρέσει η χρονιά που τελειώνει, θα λατρέψετε αυτή που έρχεται. Ευχαριστώ επίσης τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Και αν μπορείτε να μείνετε λίγα λεπτά παραπάνω, ούτω ώστε να αναφερθούμε στο πρόγραμμα της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί στη Σικελία.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

it compromise I was saying earlier when you were talking that it compromises our position and frankly the value of meeting everybody at the same time um restricts hugely what we would achieve from it. So I support your view. Peut-être pouvons-nous faire une différence entre les autorités italiennes et les acteurs qui dépendent du Parlement européen